Bene. Καλημέρα σας, αρχίζουμε. Με τις εργασίες μας η κυρία Μέρκης θα λάβει το λόγο σε σχέση με τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Έχετε λόγο κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας ε, για τη σημερινή συνεδρίαση. Σε σχέση με τις ραντιενεργές ουσίες λοιπόν, ε, ασχολήθηκα με το θέμα και λυπάμαι ιδιαίτερα διότι η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή θέλει να εντάξει αυτές τις ουσίες υπό τη συνθήκη Ευρατόμ και αν γίνει κάτι τέτοιο τότε δεν εποπτεύονται και δεν ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνεπώς θα έχουμε ένα πολύ περιορισμένο ε, ρόλο στην εποπτεία τους και δεν θα υπάρχει και δημοκρατικός έλεγχος. Η δημόσια υγεία αφορά όλους τους πολίτες, άρα μας αφορά άμεσα, γιατί εκπροσωπούμε άμεσα τους πολίτες και την υγεία τους. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον καθορισμό και αναθεώρηση της οδηγίας σε σχέση με την ε, εφαρμογή. Επειδή μιλάμε για ραδιενεργές ουσίες που εντάσσονται στην ανθρώπινη κατανάλωση, δηλαδή στο πόσιμο νερό, νομίζω ότι εντασσόμενες σε αυτή την οδηγία περιποσίμου νερού θα πρέπει να την χάνουν και τις εποπτείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλές συναφείς οδηγίες και επειδή οι ραδιενεργές ουσίες πρέπει να εντάσσονται στην οδηγία περί νερού, εάν ενταχθούν σε μια διαφορετική συνθήκη, τότε δεν εμπίπτουν στην συνθήκη περί Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι θέλουμε απλούστευση και διαφάνεια. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, δεχτεί τη συμμόρφωση με την οδηγία περί ποσίμου νερού και άλλα ύδατα όπως τον υδροφόρο ορίζοντα που δεν θα εμπεριέχει ραδιενεργές ουσίες. Επίσης, το νερό εμπεριέχεται και στη βιομηχανία τροφίμων και ε, στα τρόφιμα. Το ραδόνιο νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε σε τι ποσοστή αναλογία εμπεριέχεται στο νερό και να δούμε ποια είναι η παραμετρική του τιμή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε επαρκείς πληροφορίες ως προς το πόσιμο νερό και γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξέρουν ποια, ποιες ραδιενεργές ουσίες εμπεριέχονται στο πόσιμο νερό, όπως ορίζει και η οδηγία Περιποσίμου νερού. Εάν ε, δεν γίνει κάτι τέτοιο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποκαταστήσουν την, ε, την ποιότητα του ποσίμου νερού για να εξασφαλίσουν την υγεία των πολιτών και νομίζω ότι κάθε πέντε χρόνια θα πρέπει η Επιτροπή να αναθεωρεί τα παραρτήματα με βάση τις ε, τεχνικές εξελίξεις. Θα ήθελα να δω τι θα μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς εμείς ως πολίτες μπορούμε να ασχοληθούμε καλύτερα με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας για να εξασφαλίσουμε την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την έκθεση της κυρίας Μέρκης, θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερος ε, το μεγάλο δυναμισμό της ε, εισηγήτριας και την ενέργεια που αφιερώνει στο θέμα αυτό των ραδιενεργών ουσιών στο πόσιμο είδωρ. Πολλές από τις προτάσεις της κυρίας Μέρκης νομίζω ότι είναι περιτές. Γιατί στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε και με το αρχικό κείμενο, χωρίς τις ε, επιπλέον προσθήκες της κυρίας Μέρκης. Υπάρχουν όπως κάποια σημεία που με βρίσκουν σύμφωνο. θα πρότεινα στην τροπολογία 7 για το άρθρο 2 να συμφωνήσουμε γιατί είναι χρήσιμο να έχουμε ορισμούς. Αντίθετα, είμαι κατά της τροπολογίας 9. Κατά τη γνώμη μου είναι περίτη, για να μην πω ότι είναι και παραπλανητική. Το ίδιο ισχύει για την τροπολογία 11. Δεν με βρίσκει σύμφωνο. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να συγχαίουμε στο ίδιο κείμενο νομοθετικά κείμενα που στηρίζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις. Θα δημιουργήσει σύγχυση Θα υποβάλω πάντως και τις δικές μου τροπολογίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Χόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ και καλωσορίζω την πρόταση της κυρίας Μέρκης. Συμφωνώ ότι είναι κρίμα που ένα τόσο σημαντικό θέμα για την δημόσια υγεία, για την ανθρώπινη υγεία, να εμπίπτει στη συνθήκη Ευρατών και να μην υπάγεται στη διαδικασία συναπόφασης. Είναι πραγματικά απογοητευτικό αυτό. Μια και η οδηγία αυτή έχει άμεσες συνέπειες ε, στην υγεία των πολιτών που εκπροσωπούμε εμείς. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια συνέπεια και συνοχή, καθώς και ομοιόμορφη εφαρμογή των κριτηρίων ε, της οδηγίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πιο αυστηρή και πιο αποφασιστική, προκειμένου να εξασφαλίσει συμμόρφωση των κρατών μελών και σωστή εφαρμογή των ε, διατάξεων και αυτής της οδηγίας ε, και της οδηγίας για το πόσιμο είδωρ που ανήκει στο κεκτημένο. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι το νερό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων θα πρέπει να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογή τη συγκεκριμένη οδηγία. Η μόλυση από ραδιενέργεια, από ραδιενεργά υλικά, είναι πολύ διαφορετική από την μόλιση που συνήθως μας προβληματίζει για τα τρόφιμα, δηλαδή από βακτηρίδια, σαλμονέλα και ούτω καθεξής. Τέτοιου είδους α, ε, μολύνσεις μπορούν να αποφευθούν με ε, χρήση θερμότητας. Ε, με το βρασμό, για παράδειγμα, τα βακτηρίδια εξουδετερώνονται. Κάτι που δεν ισχύει με τα ραδιονοργά υλικά. Γι' αυτό και θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το νερό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων να πληρεί τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές με το πόσιμο είδωρ. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη στην οδηγία όχι μόνο ε, η βραχυπρόθεσμη έκθεση, αλλά και η μακροπρόθεσμη, η επανειλημμένη έκθεση σε τέτοια υλικά, γιατί η συστηματική μακροπρόθεσμη έκθεση μπορεί να ε, έχει πολύ αρνητικές συνέπειες, ε, γιατί η έκθεση γίνεται για πολύ μεγάλο χρόνο, σε ραδιενεργά υλικά και έχει σωρευτικό αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση, την ενημέρωση του κοινού, δεν αναφέρονται και πολλά στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφάνεια, ενώ πιστεύω ότι η διαφάνεια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού των πολιτών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του νερού που καταναλώνουν. Και αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνει και την ασφάλεια ότι δεν ε, περιέχονται στο πόσιμο νερό ραδιενεργά υλικά. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε τις διατάξεις για την μη συμμόρφωση. Εγώ θα προτιμούσα να θεσπιστεί η προϋπόθεση ότι σε περίπτωση μόλυσης ε, του υδροδοτικού δικτύου θα πρέπει τα κράτη-μέλη κατεπηγόντως να υποχρεούνται να εξασφαλίσουν εναλλακτική υδροδότηση δεν αρκεί να λαμβάνουμε υπόψη, να λαμβάνουμε γνώση του επίπεδου μόλι από ραδιενεργία ουσία. θα πρέπει να αποκατασταθεί η σωστή υδροδότηση και να διορθωθεί η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, συμφωνώ με τα σχόλια της εισηγήτριας και πιστεύω ότι θα πρέπει η έκθεσή μας να είναι όσο πιο έντονη γίνεται, πιο αποφασιστική και να επιμείνουμε ότι το ζήτημα αυτό είναι κέριο για τη δημόσια υγεία και δεν αφορά απλώς κάποιες τεχνικές προδιαγραφές ε, της συνθήκης Ευρατόμ. Είναι πραγματικά λυπηρό που δεν υπόκειται και το θέμα αυτό στη διαδικασία συναπόφασης. Ευχαριστώ. Νομίζω, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Κέστον Γιάνσεν, είμαι επικεφαλής της Μονάδας Προστασίας από τη Ραδιενέργεια. Καταρχάς, ευχαριστώ την εισηγήτρια και την εκτίμησή μου για την ε, πολύ καλή εργασία της εισηγήτριας και τους ε, άλλους ευρωβουλευτές που εξέφρασαν την άποψή τους. Τι απόψει αυτέ, τι αυτές ε, θεωρώ σημαντικέ είναι σημαντικό να εγκριθεί αυτή η οδηγία διότι καθεύδει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα προτείνεται υπό τη συνθήκη Ευρατών γιατί νομίζουμε ότι αυτή είναι η σωστή νομική βάση ξέρουμε τις επιπτώσεις ε, μιας τέτοιας νομικής βάσης και στις περαιτέρω συζητήσεις μας με το Συμβούλιο θα λάβουμε υπόψη τις τροπολογίες που προτείνει το Κοινοβούλιο επ' αυτού. Γενικά νομίζω ότι όλες οι τροπολογίες που προτείνει η συγγήτρια είναι στο πνεύμα της ε, πρότασής μας, ενισχύουν μερικές ε, αιτιολογικές αναφορές, ε, αιτιολογικές σκέψεις καλύτερα. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι σωστή και η διατύπωση, αν είναι κατάλληλη η διατύπωση. Διότι, ξέρετε, προσπαθήσαμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό να χρησιμοποιήσουμε την ίδια διατύπωση με την οδηγία ΕΟΚ 1998 για να μην υπάρξει καμία σύγχυση όσον αφορά τις προϋποθέσεις. Καλώς ορίζω τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν και που θέλουν να αναφερθεί σαφώς το νερό που χρησιμοποιείται στην ε, επεξεργασία των τροφίμων από τη βιομηχανία τροφίμων δεν είναι ε, αντίθετη με το πνεύμα μας γιατί είχαμε συμπεριλάβει στις αναφορές μας όλες τις ε, εξαιρέσεις που έβλεπε η οδηγία, στο άρθρο 7 συγκεκριμένα. Μιλάμε για το χώρο δειγματοληψίας όταν αφορά το νερό που χρησιμοποιεί η βιομηχανία τροφίμων, ο κλάδος ε, των τροφίμων γιατί λοιπόν να μην βάλουμε σαφώς και τον ορισμό εκπεφρασμένα. Έχω κάποιες ε, επιφυλάξεις όσον αφορά το άρθρο 9, όπως και το 4.1, όπου χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις χωρίς καμία ε, χωρίς να περιέχει καθόλου ραδιενεργές ουσίες που να προκαλούν βλάβη στην ε, ε, ανθρώπινη υγεία. Ποτέ δεν είναι εντελώς χωρίς κάποια ρεδενεργά στοιχεία ένα υλικό, οποιοδήποτε. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πού είναι τα όρια. Αναφέρεται ότι πρέπει να λαμβάνονται αμέσως, μέτρα εάν ε, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση. Βεβαίως είναι στο πνεύμα και της δικής μας, αλλά Προσπαθούμε να τηρήσουμε τη διατύπωση του 98 που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ενδεικτικές παράμετροι εάν για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί απευθείας. Και όπως ξέρετε είναι η ραδινεργός μόλυνση ε, κυρίως προκαλεί προβλήματα στην υγεία για λόγους σωρευτικούς, δηλαδή μετά από μακροχρόνια έκθεση, άρα δεν είναι θέμα να υπάρξουν αμέσως μέτρα. Χαιρετίζουμε βεβαίως ε, και την κλίση για διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων. Έχουμε ούτως ή άλλως και στη συνθήκη για την Ένωση το άρθρο 36 που καλεί τα κράτη-μέλη να κάνουν τακτικά εκθέσεις Υπάρχει λοιπόν νομική βάση για να γίνεται υποβολή εκθέσεων σε τακτικά χρονικά διαστήματα και βεβαίως είμαστε υπέρ του να υπάρχουν επαρκείς ε, εγκαταστάσεις για να γίνεται αυτό. Επίσης υπάρχει αναφορά στην οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια του 2009. Δεν είναι σωστό να αναφερθούμε σε αυτή την οδηγία, διότι αυτή η οδηγία αφορά μόνο την ασφάλεια των ε, πυρηνικών εγκαταστάσεων, ενώ η φυσική και τεχνητή ραδιενέργεια προέρχεται από πολλές αιτίε. Αν αναφερθούμε λοιπόν πιο έντονα στα άρθρα 35 και 36 της Συνθήκης Ευρατών, νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι ορθό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει η συγγήτρια. Uh, uh, Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι υπάρχει διχογνωμία επί ορισμένων θεμάτων. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε το όλο θέμα για να δούμε κατά πόσο μπορεί να επέλθει συμβιβασμός ή κατά πόσο θα κινηθούμε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χόλ για την υποστήριξή σας ως προς την κατεύθυνση που θα κινηθούμε γιατί η ανθρώπινη υγεία θα πρέπει να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής αυτής της γνωμοδότησης και όλα τα συναφή θέματα μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής ΕΜΒΗ ή όταν μιλάμε για θέματα που άπτονται της πυρηνικής ασφάλειας. Τώρα, ως προς τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει διαφορά απόψεων σε σχέση με τη νομική βάση. Εγώ τάχθηκα σαφώς υπέρ της Ένωσης σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό και να το εντάξουμε στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή πρωτίστως και όχι της Ευρατών. Εσείς θεωρείτε ότι η σωστή βάση είναι η Ευρατών. Θα πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ μας και θα επανέλθουμε επί του θέματος. Σας ευχαριστώ ως προς την ε, υποστήριξή σας για την, ε, ως προς τη βιομηχανία τροφίμων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε, να έχουμε πιο σαφή θέση επί του θέματος. Υπάρχει επιφύλαξη ως προς τη συμπερίληψη ορισμένων άρθρων από εσάς έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθόλου ραδιενεργές ουσίες ε, Καταλαβαίνω την επιφύλαξή της ως προς τη χρήση της λέξης free, δηλαδή ελεύθερες ή ελεύθερα από ραδιενεργές ουσίες. Θα το δούμε ως προς τη διατύπωση. Ως προς την ποιότητα του νερού, θα ήθελα να επανέλθω στη συνθήκη Ευρατόμ. Η ποιότητα του νερού εντάσσεται στη συνθήκη της Λισαβόνας, σαφέστατα. Επειδή εντάσσουμε και την πυρηνική πτυχή, θέλετε να ενταχθούν όλα στην Ευρατόμ. Τι έχει μεγαλύτερη σημασία, ποιο σκέλος έχει μεγαλύτερη σημασία, η ανθρώπινη υγεία, το πόσιμο νερό, η ποιότητα του πόσιμου νερού ή η πυρηνική πτυχή του θέματος, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι βαρύνει περισσότερο και προς τα εκεί να κινηθούμε. Για μένα είναι σαφές ότι η ανθρώπινη υγεία είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο του θέματος και της γνωμοδότησης αυτής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια, την κυρία Μέρκης. Ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 3η 11 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο επόμενο θέμα με εισηγητή τον κύριο Λάγκεν, ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Έχετε το λόγο κύριε Λάγκεν. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, που θα αποστείλει η Επιτροπή Έρευνας για την έκθεση Ζουβάν στην ΙΜΚΟ. Μετά από 10 χρόνια συζητήσεων, πάνω από 10 χρόνια, η Κομισιόν προτείνει μια οδηγία για την ε, χορήγηση, την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Ήταν καιρός, κατά τη γνώμη μου, αλλά ξέρουμε ότι ορισμένοι του κλάδου την απορρίπτουν κατηγορηματικά. Συζήτησα με τον συνάδελφο Ζουβά, κοίταξα το έγγραφο εργασία του και καταλαβαίνω ότι την υποστηρίζει και αυτό είναι σωστό αλλά θα πρέπει να υποβληθούν κάποιες τροπολογίες στο υπάρχον κείμενο. Η σημασία των συμβάσεων παραχώρησης, όπως λέει και η Κομισιόν, είναι μεγάλη. Γύρω στο 60% των ε, συμβάσεων δημοσίου ιδιωτικών φορέων είναι συμβάσεις παραχώρησης. Είναι δημόσιες ε, συμβάσεις από υπηρεσίες μέχρι δημόσια έργα. Έχουμε σαφείς οδηγίες πώς πρέπει να γίνονται οι προκηρύξεις και τι διατάξεις πρέπει να ισχύουν. Για τις παραχωρήσεις όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα η Επιτροπή προτείνει μια διαδικασία με δύο στάδια. Πρώτα, να υπάρχει μια γενική υποχρέωση δημόσιας προκήρυξης όταν είναι πάνω από 5 εκατομμύρια. Αυτό βεβαίως ε, είναι κατάλληλο για τα δημόσια έργα. Αλλά για τις υπηρεσίες, ε, για συμβόλαια μεταξύ 2,5 και 5 εκατομμυρίων, προτείνει απλώς υποχρέωση δημοσίευσης. Στο δικό μου κείμενο της 28ης έκτου Καταργώ αυτή την ε, διαφοροποίηση και προτείνω η κατώτατη τιμή για τις υπηρεσίες να πάει στα 2,5 εκατομμύρια. Οπότε δεν χρειάζεται ε, αυτή η διαφοροποίηση, δημοσίευση και προκήρυξη, διαγωνισμός. Πιστεύω ότι και παραχωρήσεις, συμβάσεις παραχώρησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υπόκειται στην υποχρέωση δημοσίευσης. Βεβαίω τα κράτη-μέλη μιλάνε για μεγαλύτερα συμβόλαια, όπου ο δημόσιος ε, τομέα δεν έχει υποχρεώσει έναντι της Ευρώπης. Έχω διάφορα παραδείγματα από την ε, Ρινανία Παλατινάτο, το, την ε, χώρα μου, όπου για ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που είναι του περιφερειακού της Νιρεμβέργης δεν έγινε σωστή διαδικασία και υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη διαμάχη. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί λόγοι για να γίνει αυτή η αλλαγή και επιπλέον στις τροπολογίες μου αναφέρω ότι πρέπει να εισαχθεί αυτή η τροποποίηση στην οδηγία, δηλαδή ότι στο μέλλον τα βασικά σημεία της σύμβασης θα πρέπει να ισχύουν ακόμη και αν δεν ισχύουν τα συμβόλια, τα κατόφλια για κάθε χωριστό τμήμα, εφόσον συνολικά για τη σύμβαση το ποσό είναι πάνω από το όριο. Και αυτό θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε την έλλειψη διαφάνειας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει κενό. Ελπίζω να το δεχτεί ο συνάδελφος Ζουβά. Ο τρίτος τομέας, συνολικά, έχω υποβάλει 55 τροπολογίες, δεν τις αναφέρω βέβαια όλες. Πώς πρέπει λοιπόν να αναφέρουν κάποιες άλλες τροπολογίες μου να διευκρινίσουμε κάποιες νομικές έννοιες. Η Κομισιόν λέει ότι μπορεί να καταργηθεί η διαδικασία διότι η τιμή μπορεί να υπερβαίνει τις προδιαγραφές. Δηλαδή, Μπορεί λοιπόν ο αναθέτων να θέσει ε, αυθαίρετα μία τιμή και μετά να αποφασίζει εάν οι προσφορές είναι κατάλληλες με βάση αυτή την αρχική τιμή. Αυτό δημιουργεί δυνατότητες αυθαιρεσίας, διότι μπορεί να αφαιρέσει πρόσβαση από όλους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί. Δηλαδή, εάν η αξία υπερβαίνει από πάνω, κατά πάνω από 20% για να μην μπορεί να εξαιρέσει ο αναθέτων. Αντίστροφα, μπορεί να ε, προβλέπεται τώρα ότι μπορεί να απορριφθεί μία ε, προσφορά εάν είναι ασυνήθιστα χαμηλή. Ασυνήθιστα χαμηλή είναι ασαφές. Προτείνω λοιπόν να απορρίπτεται αν είναι πάνω από 20% κάτω από τη μέση τιμή των άλλων προσφορών. Αυτό νομίζω δίνει περισσότερη νομική ασφάλεια και λιγότερες δυνατότητε καταχρήσεων. Ένα σημείο που δημιουργεί διαμάχες είναι η λεγόμενη έννοια του πλήρους κόστους. Η Κομισιόν προτείνει να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κόστος ζωής για να υπολογιστεί το συνολικό κόστος του συμβολέου συμπεριλαμβανομένων και των ε, στοιχείων του κόστους παραγωγής και των επιπτώσεων, του κόστους των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή. Αυτά είναι ασαφή. Όλα αυτά λοιπόν τα ε, ε διαγράφω, καθώς και το κόστος παραγωγής. Εμάς μας ενδιαφέρει το τελικό προϊόν. Μας ενδιαφέρει αυτό που θα μας προτείνουν. Αλλιώ για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε όλα τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία του κόστου που αναφέρονται χρειάζεται τρομερή γραφειοκρατική σπατάλη. Επίσης ε, υπάρχουν και οι επιχειρήσεις που είναι δημοσίου δικαίου, οι εσωτερικές όπως λέγονται επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν διαγωνισμούς. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αυτές οι εσωτερικές εταιρείες Βεβαίω δεν πρέπει να απαγορεύουμε γενικά τις, ε, τη συμμετοχή τους, αλλά πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες ε, προϋποθέσεις. Δηλαδή, εάν στο παρελθόν είχαν κάνει ένα μεγάλο ποσοστό, 80% των ε, συμβάσεών τους με το δημόσιο τομέα. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου του 2006 και γι' αυτό εισάγω ένα κατώτατο όριο. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10% ε, ιδιωτική συμμετοχή. Ιδίως στον τομέα των μεταφορών, σε συγκεκριμένα κράτη, υπάρχει ένα όριο του 5% και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή ενός ανταγωνιστή αποφάσισε ότι εφόσον υπάρχει συμμετοχή έστω και ε, λίγο πάνω από το 0, δεν θεωρείται ότι αυτή η επιχείρηση πρέπει να απαγορεύεται να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς. Εγώ προτείνω να πάμε στο 10%. Το επόμενο σημείο πώς θα εξασφαλίσουμε τη διατήρηση διατάξεων δικαίου. Είναι σαφές ότι όποιες προσφορές παραβαίνουν κανόνες δικαίου, κάποιες ε, νομικές διατάξεις φυσικά πρέπει να αποκλείονται. Το θέμα όμως είναι για παράδειγμα αν υπάρχουν συγκεκριμένες συλλογικές συμβάσεις. Θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιούμε τις δημόσιες συμβάσεις για να παρεμβαίνουμε στις συλλογικές συμβάσεις ε, των εργαζομένων στις εταιρείε που κάνουν προσφορές. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να γίνεται. Ωστόσο, εάν υπάρχουν ε, σοβαρές παραβιάσεις, εάν έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν σοβαρές παραβιάσεις των κοινωνικών διατάξεων ή των περιβαλλοντικών διατάξεων. Ενώ η Κομισιόν προτείνει εάν ε, υπάρχει ενδεχόμενο τέτοιων παραβιάσεων. Αυτό είναι ασαφές. Συνολικά λοιπόν έχω ε, υποβάλει 55 τροπολογίες. Δεν ξέρω αν έχει ήδη μεταφραστεί η έκθεση, δεν την είδα. Εγώ τήρησα την προθεσμία υποβολή του κειμένου μου στις 26 και οι συνάδελφοι θα έχουν μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου προθεσμία για να υποβάλουν τροπολογίε, Η επί τη Ζουβά ε, θα ακολουθήσει μετά. Έχουμε λοιπόν ε, τη δυνατότητα να συζητήσουμε μετά τι διακοπέ για τη γνωμοδότησή μας. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι κάθε αναθέτων πρέπει να, να μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Δεν χρειάζεται να κάνει προκήρυξη. Αλλά αν υπάρχει ε, συμμετοχή ιδιωτικού φορέα, όπως γίνεται συνήθω για την παραχώρηση, τότε πρέπει να ισχύσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων, εφόσον το όριο είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Με λοιπόν, αυτές τις συνθήκες μπορεί οποιοδήποτε αναθέτων, δεν χρειάζεται βεβαίως υποχρεωτικά να συμμετάσχουν ε, ιδιωτικές εταιρείες στο έργο του, αλλά εάν πρόκειται να συμμετάσχουν τότε θα πρέπει όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν, πρέπει να είναι σαφή τα όρια, σαφή οι διατάξεις, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε, να μπορούμε επίσης να ε, ε, αμφισβητήσουμε ενώπιον των δικαστηρίων, των δικαστηρίων την διαδικασία παραχώρησης. Ευχαριστούμε τον κύριο Λάγκεν. Η κυρία Μέρκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον συνάδελφο για την εκτενή παρουσίαση που μας έκανε. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πολλά κοινά σημεία, γιατί συμμερίζομαι το στόχο σας να περιοριστεί η υπερβολική γραφειοκρατία, οι περιττές διατυπώσεις και να απλουστεύσουμε τα πράγματα όσο γίνεται. το θέμα της φρενίτιδας του διοξιδίου του άνθρακα που έχει πάθει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν είμαι κατά αυτής της φρενίτιδας. Θα το εξετάσω βέβαια μετά την παρατήρηση που κάνατε, ενδελεχέστερα. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γόνιμη συζήτηση για το θέμα αυτό. Για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια χρυσή τομή ή αν θα εμείνουμε ο καθένας στις θέσεις του. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της οδηγίας, νομίζω ότι την περιμέναμε εδώ και καιρό. Δεν είμαι κατά της ιδέας της οδηγίας αυτής για ένα τέτοιο θέμα. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για τις παραχωρήσεις και μετά από ένα κατόφλι οι παραχωρήσει μπορεί να επηρεάσουν την ε, νέα αγορά και άρα θα πρέπει να υπόκεινται στην κοινοτική νομοθεσία. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προβλέψει κάποιε διακιστικέ προποθέσει και διευκρινήσει για να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση στην αγορά των παραχωρήσεων και στους διάφορου διαγωνισμού. Βέβαια, συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε ελαστικότητα. Θα πρέπει να καλυφθούν κάποια διαδικαστικά θέματα, ώστε το πεδίο εφαρμογή των παραχωρήσεων να προσδιορίζεται σαφώ. Το λάθος όμως που συνήθως διαπράττει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι είμαστε υπερβολικά σχολαστικοί και διεξοδικοί για τον τρόπο, αντί να είμαστε πιο σχολαστικοί ως προς το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ε, θα πρέπει να χαράξουμε το στόχο, το αποτέλεσμα με λεπτομέρειες, αλλά να αφήσουμε πιο χαλαρές τις διαδικασίες και πιο γενικές. Δεν θα πρέπει ε, να επιφέρουμε μεγάλη γραφειοκρατία και περιπλοκή στη διαδικασία, γιατί οι τοπικέ και οι περιφερειακές αρχές αυτό φοβούνται, ότι η οδηγία θα περιπλέξει τα πράγματα, γιατί το ίδιο πρόβλημα έχουμε με την οδηγία για τι δημόσιες προμήθειες. Η οδηγία αυτή λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στα κύριο θέματα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης ε, θέσπισης πολιτικών, αλλά με το στόχο της νομικής ασφάλειας και της ομοιομορφίας για τον τρόπο δημοσίευση μιας ε, σύμβασης, τον τόπο και το χρονικό πλαίσιο. Μια άλλη σημαντική παρατήρηση για την έκθεση του κυρίου Λάγκεν είναι ότι υπάρχουν κάποιες αφιβολίες για το κατά πόσο θα πρέπει να μειώσουμε το κατόφλι των παραχωρήσεων από τα 5 εκατομμύρια στα 2,5 εκατομμύρια. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας μείωσης. Η επίπτωση της παραχώρησης στην εσωτερική αγορά εξαρτάται και από τη διάρκεια της. Και συναφέ θέμα είναι μια πολιτική που θα είναι φιλική προ τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, Πολλά λέγονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω τη κρίση, και είναι σωστό. Αν έχουμε υψηλό κατόφλι λοιπόν θα υπάρξουν περισσότερε παραχωρήσει χωρί ε, ε, διαγωνισμού και μια πολιτική πολύ πιο φιλική προ τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, προτιμώ να διατηρήσουμε τα 5 εκατομμύρια ω κατόφλι. Και τέλο. για τον έλεγχο ε, και για το κατά πόσο υπάρχει αρκετή ελαστικότητα ε, ώστε οι δημόσιες αρχές να θεσπίσουν ε, σημαντικά κατά τη γνώμη τους ειδικά κριτήρια. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και τροποποίηση ενό τμήματο των παραχωρήσεων. Αναφέρεται 5% τη συνολική αξία ω επιτρεπόμενο όριο για τι αλλαγέ. Δεν ξέρω όμω αν είναι αρκετά ελαστικό αυτό το ποσοστό το δικό μας ε, μάντρα, το δικό μας ε, σύνθημα είναι ελαστικότητα και πάλι ελαστικότητα. Και αυτό το σημείο θα πρέπει να το επισημάνομαι ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Λιζόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την, την Επιτροπή, για την συνολική της υποστήριξη, για την ύπαρξη οδηγίας. Δεν θα ήθελα να θίξω όλα τα επιμέρους ζητήματα. Θα ήθελα όμως να πω ότι όσον αφορά τα κατόφλια, και ευχαριστώ τον εισηγητή, λαμβάνω υπόψη την ιδέα του εισηγητή, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε ανώτερα κατόφλια, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη ένα ελεγχόμενο λογικό κόστος μέσα στα πλαίσια του επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. Και βεβαίως θέλουμε να υπάρχει νομική ασφάλεια, δηλαδή να υπάρχει μία ενιαία τιμή, μία ενιαία αξία και απλούστευση. Εάν υπήρχαν διαφοριακές ε, οριακές τιμές σε σχέση με τα, τους δύο τύπους παραχωρήσεων, θα σήμαινε ότι οι δημόσιοι φορείς θα βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση γιατί θα επρόκειτο για μία παραχώρηση υπηρεσιών, αλλά θα την παρουσίαζαν ως παραχώρηση έργου. Ε, έτσι ώστε να μπορούν να κινηθούν κάτω από τα 5 εκατομμύρια. Γιατί στην ουσία θα επρόκειτο για παραχώρηση υπηρεσίας και όχι παραχώρηση έργου και θα μπορούσε να ενταχθεί αλλού. Πέρα από τα κατόφλια θα ήθελα να δούμε και το πεδίο εφαρμογής, ε, δηλαδή λάβαμε υπόψη τον ορισμό της παραχώρησης που θα πρέπει να βελτιωθεί και να αποσαφινιστεί και μας ε, απασχολεί το θέμα. Το εξετάζουμε δηλαδή. Σε σχέση με τα άλλα ε, ζητήματα που εφήγησαν, δηλαδή επιπρόσθετους αποκλισμούς, λαμβάνοντας υπόψη το εργατικό δίκαιο, τα περιφαλλοντικά και άλλα ζητήματα, ως προς την παραχώρηση, ως προς παραχωρήσεις και τις τροποποιήσεις παραχωρήσεων, καθώς και την ιδιωτική συμμετοχή που θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή σε επίπεδο 10%. Όλα αυτά συζητήθηκαν μέσα στα πλαίσια των δημόσιων συμβάσεων και θα δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή των δημοσίων συμβάσεων για να ενταχθεί και αυτή η πρόταση περί παραχωρήσεων. Επίσης, θα ήθελα να σας τονίσω ότι οι απόψει σας θα ληφθούν επαρκώς υπόψη και συνεργαζόμαστε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα κοινό αποδεκτό κείμενο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω το εξής. Ήδη συνέβη χτες και επαναλαμβάνεται και σήμερα. Δηλαδή ένα συνάδελφος ζητά το λόγο αφού παρέμβει η Επιτροπή. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο κύριος Μενίν μπορεί να παρέμβει για ένα λεπτό, αλλά δεν θα ήθελα. Ο κύριος Ένα θα παρέμβει τώρα, αλλά δεν θα ήθελα να επαναληφθεί αυτό, διότι δεν είναι η τρέχουσα διαδικασία και δεν είναι σωστό. Ζήτω συγγνώμη. Ε, αποκλεισμοί για ε, λόγους μη σεβασμού του εργατικού και κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρόσθετα να συμπεριλάβουμε τους υπεργολάβους. Γιατί πολύ συχνά ο, ε, αυτός που έχει αναλάβει τη σύμβαση βάζει τους υπεργολάβους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και δεν ε, καταδικάζεται ποτέ κανείς. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Εξήγησα μόνο ορισμένε από τι τροπολογίε, αλλά μπορείτε να τι διαβάσετε. Έχω υποβάλει και τροπολογίε για το ύψο των υπεργολάβων, που φυσικά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Τώρα, ποιε είναι οι ελάχιστε τιμέ, πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ μα ε, ιδιαίτερα. Άλλαξα το κατώτατο όριο για την κατάσταση μεταξύ 2,5 και 5 στα άρθρα 27-28 δηλαδή να προβλέπεται, να προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης. Δηλαδή θα αλλάξουμε την τιμή ή θα αλλάξουμε τη διαδικασία. Βεβαίως, το λέω στην ε, σοσιαλδημοκράτη συνάδελφο, βεβαίως για να συμπεριλάβουμε το συνολικό κόστος πρέπει να έχουμε τάξη μεγέθους που να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Και εδώ θα βρούμε λύση πιστεύω. Κατά τα άλλα και, εσύ, και εσείς νομίζω έχετε την φιλοδοξία αυτό που θα αποφασίσουμε να βοηθήσει την ε, επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή και όχι να μπει απλώς, απλώς ως παράδειγμα. Στόχος μου λοιπόν είναι η γνωμοδότησή μας να μπορέσει να τη χρησιμοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή. Ευχαριστώ και με χαρά θα συζητήσω τις τοπολογίες που θα το Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Όπως ήδη ελέγχθη, οι τροπολογίες πρέπει να ενταχθούν, να υποβληθούν, με μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στις 12. Διακόπτουμε για τρία λεπτά. Bene, Μπορούμε να επαναλάβουμε, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Περιμένω να καθίσετε όλοι. Allora, passiamo ai voti. Περνάμε στη σημερινή μας ψηφοφορία. Το πρώτο θέμα είναι η ενεργειακή απόδοση ψηφίζουμε το κείμενο ως έχει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ψηφίσατε όλοι. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία γιατί Δημιουργήθηκαν μερικά προβλήματα με τις κάρτες σας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 42 υπέρ. 42 ουδής κατά και δύο αποχές. Πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εκιούζα. Πέρας. 42 υπέρ, ουδής κατά, Δύο αποχές. Εγκρίνεται το κείμενο. Να συγχαρούμε τον εισηγητή και την Επιτροπή για το έργο της. Allora, passiamo al Επόμενο θέμα, επόμενη ψηφοφορία. Συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συμβουλίου για τον έρασμο για όλους. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας γίνει μία επαλήθευση. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 30 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται η 52. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 και 3 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές ε, φαίνεται ότι έχει απορριφθεί αλλά σε ελέγξουμε την 8 παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ισοψηφία άρα απορρίπτεται 23 προς 23. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφίας. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ο συμβιβασμός. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβιβασμού 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 με την προφορική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ, με την προφορική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε την, ε, την 15. Ε, την 15. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται πράγματι. Με 27 ψήφους, 80 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 80... θέλετε να ελέγξουμε, ας ελέγξουμε την 83, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Η κυρία Νίμπλερ. Δυστυχώς έχω ξεχάσει την κάρτα μου και είμαι και εγώ υπέρ, παρακαλώ σημειώστε. Εγκρίνεται 25 έναντι 22 εγκρίνεται. Ογδόντα τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε, εντάξει. Ας ελέγξουμε την 89, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 18 έναντι 27 απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 23, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας για την 23 εγκρίνεται. 25 έναντι 20. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 με την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά αποχές μου φαίνεται ότι έχει απορριφθεί, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Η ισοψηφία 23 προς 23 η κυρία Νίμπλε απορρίπτεται. Είναι πιο σίγουρο το αποτέλεσμα, δεν έχουμε ισοψηφία. 24 ψήφοι κατά με την κυρία Νίμπλερ. 28 υπέρ. Όχι, κάνε, κάνω λάθος, με συγχωρείτε. 93, 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 95 με την προφορική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά ας ε, ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται με ισοψηφία, λέει η Πρόεδρος. Όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται. 26 υπέρ, 21 κατά. 31 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά. Αποχές ε, νομίζω πρέπει να επαληθεύσουμε, δεν είναι απόλυτα σαφές. 33 επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Όπως και πριν, 27 εναντί 20 εγκρίνεται, 96. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε, ελέγχουμε λέει η πρόεδρος, δεν γίνεται διαφορετικά. 96, 96. 96. Απορρίπτεται. 20 έναντι 27. Κατά. 97 με την προφορική. Υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε και πάλι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αλλάζεται, αλλάζουν γνώμη πολύ από ό,τι φαίνεται. Οπότε καλύτερα να ελέγξουμε. Πέρας. 25 έναντι 22, άρα εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 98. Πέρας. Η κυρία Νίμπλερ απορρίπτεται. Ισοψηφία 24 υπέρ, 24 κατά. Καταψήφισε η κυρία Νίμπλερ αυτή τη φορά. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε, ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 36, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. 26 υπέρ, 19 κατά, 20 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε. Την 37 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ, 21 κατά. Η κυρία Νίμπλερ διαθέτει πλέον την κάρτα της. 27-20, άρα εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Α, με συγχωρείτε, εγκρίνεται, λέει η πρόεδρος. Κατά τη γνώμη μου εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται 27 έναντι 21. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση 41 υπέρ 4 κατά αποχές να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Πέρας της ψηφοφορίας να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Και περνάμε στην έκθεση Τζαβέλα για τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050. Δύο λεπτά διάλειμμα διακοπή για όσους θέλουν, για όσους θέλουν να αποχωρήσουν. Complimenti Turmes. Ciao. Bene. La parola alla collega Zavella. Η κυρία Τζαβέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, σε αυτή τη φάση της έκθεσης σε αυτή τη φάση της έκθεσης δεν θα ήθελα να πάρω το χρόνο Okay. Δεν θα ήθελα να πάρω το χρόνο από τους συναδέλφους μου. Σας έχει κοινοποιηθεί το σχέδιο της εκθέσεως και αυτή τη στιγμή σας δίνω και ένα συνημένο σημείωμα με τροπολογίες τις οποίες θα πρότεινα να υποβάλαμε όλοι μαζί. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και το συνεργάτη μου τον Κωνσταντίνο τον Λεβογιάννη για τη βοήθεια που μου παρήχανε στη σύνταξη αυτού του σχεδίου έκθεσης. Ε, δεν θα πω τίποτα άλλο κυρία Πρόεδρε, προτιμώ να ακούσω τι θα πούν οι συνάδελφοί μου επί του σχεδίου το οποίο τους έχω υποβάλει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν κατάλαβα τι είπατε γιατί δεν είχα ανοιχτό το ακουστικό σα. Λοιπόν, έχω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Τζαβέλα για την έκθεση. Πολύ καλή βάση για τη συζήτηση. Είναι και η δυνατότητα, μου δίνει και η δυνατότητα να ευχαριστήσω και την Κομισιόν. Αντίθετα με πολλά έγγραφα που διάβασα τα τελευταία χρόνια, επιτέλους μας υπέβαλε ένα κείμενο που βοηθάει τη συζήτηση. Δηλαδή προσπαθεί να παρουσιάσει τα διάφορα σενάρια, να μας δώσει τη βάση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις, να διαλέξουμε μεταξύ των εναλλακτικών ε, δυνατοτήτων. Όχι να μας δίνει στόχους, στόχους, στόχους, στόχους, στόχους, ούτως ώστε και η οικονομία και η πολιτική και οι απλοί άνθρωποι να μην μπορούν να καταλάβουν. Μας δίνει τις εναλλακτικές λύσεις. Μπορούμε να δούμε αν συμφωνούμε που είναι πλήρης η παρουσία ενός σεναρίου ή που χρειάζεται επιπλέον διευκρίνηση. Πολύ σωστή λοιπόν μέθοδος εργασίας και ευχαριστώ για αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Και η έκθεση είναι πολύ σωστή γιατί αναφέρεται σε σημεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Τζαβέλα ότι η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια του εφοδιασμού είναι τα δύο βασικά θέματα στον ενεργειακό τομέα. Συνολικά αυτόν τον χάρτη πορείας θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε ως ευκαιρία, ούτως ώστε να διευκρινίσουμε, εάν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στους βασικούς στόχους και από εκεί μετά να βγάλουμε και τις επιπτώσεις γιατί στο παρελθόν είχαμε το πρόβλημα ότι θέταμε πολλούς στόχους παράλληλα και τα μέτρα μετά που λαμβάναμε βάση αυτούς τους στόχους ήταν αντιφατικά το ένα προς το άλλο. Δεν επιτύχαμε πολλά γιατί ε, προσπαθούσαμε να προωθήσουμε πολλούς και πολύ διαφορετικούς στόχους την ίδια στιγμή. Εάν στόχος για παράδειγμα, και πρέπει να συμφωνήσουμε, εάν θα συμφωνήσουμε ότι στόχος μας ε, είναι οι στόχοι για το διοξείδιο του άνθρακα, μετά θα δούμε πώς θα οδεύσουμε προς αυτόν τον στόχο χρόνο το χρόνο. Αλλά επίσης πρέπει να συζητήσουμε και είναι τμήμα της έκθεσης να συζητήσουμε ειλικρινά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές οδοί, διαφορετικά μέσα για να καταλήξουμε στους στόχους μας για το διοξείδιο του άνθρακα. Η έκθεση το αναφέρει σαφώς. Λέει, δεν αποφασίζουμε εμείς ως Ευρώπη, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν τι ενεργειακό μείγμα θέλουν να έχουν. Και αν ο στόχος μας είναι το διοξείδιο του άνθρακα, αν είναι τόσο σημαντικό, αν θέλουμε να τον θέσουμε ως πρώτη προτεραιότητα, τότε πρέπει να δούμε ποιε πηγέ ενέργεια θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχου μας περισσότερο ή λιγότερο. Δεύτερον, η επιβάρηση της βιομηχανίας, η ενεργειακή απόδοση, το κόστος είναι επίση σημαντικοί παράγοντε Τον τελευταίο καιρό πρέπει να εξετάσουμε με τι τρόπο θα βοηθήσουμε την οικονομία μας για να υπάρξει ανάπτυξη. Άρα τα μέτρα που λαμβάνουμε στον ενεργειακό τομέα έχουν επιπτώσεις και εδώ. Τι επιπτώσεις θα έχουν. Τι θεωρούμε σκόπιμο. Τι θεωρούμε ευφυές. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε και για τις δυνατότητες των ανανεωσίμων. Υπάρχουν ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν. Πώς θα εξαγάγουμε το μέγιστο από αυτές τις πηγές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αρκετά πιστεύω ότι ε, ε, πιστεύω λοιπόν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι η καλύτερη μέθοδος που χρησιμοποιούν διάφορα κράτη-μέλη για τις ανανεώσιμες. Θέλουμε υψηλότερη απόδοση. Η Κομισιόν εδώ και χρόνια μας έχει πει δεν θα ήταν πιο ευφυές να συζητήσουμε τις ανανεώσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα επανέλθω σε αυτό. Αλλά όλα αυτά είναι τμήματα του χάρτη πορείας. Πρέπει να εξετάσουμε. Με ποια μέσα, με ποια εργαλεία θα επιτύχουμε τους στόχους που θεωρούμε σημαντικούς. Και γι' αυτό θεωρώ πως είναι πολύ καλή αυτή η προσέγγιση. Και ευχαριστώ πολύ Έχουμε μιλήσει και για το σχιστο, σχιστολιθικό αέριο. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι πολύ δύσκολη η εξόριξη, η εκμετάλλευσή του. Αλλά αν έχουμε τέτοιε ανάγκε ενέργεια. και αν δεν θέλουμε να είμαστε εξαρτημένοι από άλλου, πρέπει να σκεφτούμε. Εάν τι πηγέ που ήδη έχουμε, για παράδειγμα, με το σχιστολιθικό, δεν θα πρέπει να τι αξιοποιήσουμε. Δεν υπάρχει τρόπο να τι αξιοποιήσουμε χωρί να επιβαρύνουμε το κλίμα και το περιβάλλον σε απαράδεκτο βαθμό. Εμεί δεν λέμε ότι δεν γίνεται, λέμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Θα πρέπει να δούμε και τι ευκαιρίε έχουμε από του κινδύνου. Σωστό επίση, αν μα ενδιαφέρει η ε, ασφάλεια εφοδιασμού, πρέπει να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τον άνθρακα. Αν όμω το πιο σημαντικό για μα είναι το διοξείδιο του άνθρακα, τότε να ε, εξετάσουμε πώς θα περάσουμε σε μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας ε, δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα. Όλα συσχετίζονται. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα που μας δίνονται οι εναλλακτικέ. Και στο κέντρο της προσοχής μας είναι τα δεδομένα. Ίσως λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να επιτύχουμε συνένεση. Η δουλειά μας δεν είναι το ε, καλύτερο δυνατό, το σημαντικό είναι πώς θα επιτύχουμε το ταχύτερο, με το μικρό δυνατό κόστος, αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τζαβέλα για την ήδη επιτελεστή εργασία και προσβλέπω σε περαιτέρω καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ehm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της. Η έκθεση της είναι πολύ συγκροτημένη και μας δίνει μια καλή επισκόπηση των βασικών σημείων σε αυτό το χάρτη πορείας. Έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Όντως η έκθεση αυτή είναι μεστή, συγκροτημένη, αλλά δεν είναι αρκετά πλήρης, ε, δεν ε, καλύπτει όλες μας τις ε, επιθυμίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει μία σειρά προτάσεων και σενάριων και είναι ενδιαφέρουσε οι πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μειονέκτημα αυτής της πρότασης, και αυτό θα πρέπει να το διορθώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ότι δεν λαμβάνει μία απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν εκφράζει προτιμήσεις, ενώ θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο χωρίς να σφετερίζεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, αλλά λέγοντας τουλάχιστον ποιος είναι ο κοινό στόχος. Θέλουμε μια ασφάλεια στην αγορά. Σε τι θα επενδύσουμε, τι επενδύσεις θα αποφύγουμε, ποιες είναι οι τεχνολογίες του μέλλοντος. Και ποιες τεχνολογίες θέλουμε να υποστηρίξουμε. Και αυτό θα επισημάνω στην τροπολογία μου. Θέλουμε πιο συγκεκριμένους και πλήρεις στόχους ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να σας θα δώσω και μερικά παραδείγματα. Στην παράγραφο 3 πολύ σωστά ε, αναφέρεται τη συνάφεια μεταξύ της ενέργειας και της επιλογής των μελλοντικών ενεργειακών συστημάτων. Λέτε ότι έτσι θα διέλθουμε από την κρίση εξασφαλίζοντας μία αηφορία της ανταγωνιστικότητάς μας. Και πολύ εύστοχα μας λέτε ότι οι στόχοι της ε, Ευρώπης 2020 θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά και να υπάρχει και έλεγχος της εφαρμογής τους και επίση να τεθούν ε, νέοι στόχοι μέχρι το 2030. Αλλά θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο σαφείς, κυρία εισηγήτρια, και να πούμε με σαφήνεια, με λεπτομέρειες, πώς βλέπουμε εμείς τους στόχου μέχρι το 2030, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ενεργειακή απόδοση, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτά τα περιλαμβάνει ήδη η στρατηγική του 2020. Ποιες είναι όμως και οι δικές μας ε, προτεραιότητες και στόχοι. Επίσης, γιατί λέμε μόνο 2030, γιατί να μην πούμε και 2040, 2050, να υιοθετήσουμε και μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Με δύο λόγια λοιπόν, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τους στόχους μας. Αυτό θα πρέπει περισσότερο να εξετάσουμε και να είμαστε και φιλόδοξοι στην προσέγγισή μας. Γιατί στο παρελθόν τα θετικά στοιχεία της στρατηγικής α, ε, ε, οφείλονταν στην ε, θέσπιση σαφών στόχων Μερικέ ε, φορέ, τα κράτη-μέλη ήταν ε, πρόθυμα και επιφυλακτικά, αλλά χάρη στους συγκεκριμένους στόχους ε, ενθαρρύνθηκαν για να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. Τώρα, για το δημόσιο τομέα, παράγραφοι 5 και 17. Πολύ σημαντικό ο δημόσιο τομέα και πολύ σωστά τον υπογραμμίζεται. Χρειαζόμαστε ένα δραστήριο δημόσιο τομέα και ταυτόχρονα και αποτελεσματικό. Και αυτό φυσικά γίνεται μόνο με μια εύρυθμη και διαφανή αγορά. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά και εδώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Οι δημόσιες αρχές, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να συντονίζουν τις προσπάθειές τους και ταυτόχρονα να δραστηριοποιηθούν και να διορθώσουν και τις ατέλειες της αγοράς, τις, τις λειτουργίες της. Νομίζω ότι και αυτό το σημείο θα μπορούσε να ενταχθεί στο μελλοντικό μα όραμα. Να επικεντρωθούμε και στις υποδομές και να ζητήσουμε πιο δραστήριε δημόσιες αρχές και να τις ενθαρρύνουμε στις προσπάθειές τους. Τώρα, η λύση no regrets, ε, να μην μετανιώνουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο του χάρτη πορείας σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επενδύσουμε στην ενεργειακή απόδοση και σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. Το αποφασίσουμε και δεν υπαναχωρούμε. Είναι πολύ σημαντικό να μην υπαναχωρήσουμε. Είναι μια οριστική επιλογή και θα πρέπει να την στηρίξουμε. Ανανεώσιμες πηγέ ενέργειας. Χρειαζόμαστε, ε, επαναλαμβάνω, σαφεί στόχους, σαφώ προσδιορισμένου στόχους. Ξέρω ότι μακρηγορώ, αλλά νομίζω ότι αξίζει που και που να υπησερχόμαστε σε λεπτομέρειες και να μην ε, περιοριζόμαστε σε γενικότητες και αοριστείες. Ξέρω ότι μακρηγορώ, αλλά έχω πολλά σημεία. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικό να εξετάσουμε όχι μόνο τα μεγαλεπίβολα σχέδια, για την Βόρεια Θάλασσα, για παράδειγμα, ε, υπεράκτιες ε, ανεμογεννήτριες, αλλά να δώσουμε έμφαση και στα τοπικά προγράμματα και σχέδια. Επίσης είναι σημαντικό. Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να αναφερθεί και είμαι βέβαιη ότι θα προξενήσει και σφοδρές συζητήσεις. Το θέμα της δέσμευσης όμως και της αποθήκευσης του άνθρακα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν θα πρέπει να το αναφέρουμε έτσι γενικά και όριστα με οποιαδήποτε τεχνολογία και πάση θυσία. Χρειαζόμαστε επίσης φυσικό αέριο για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα που εκλείεται από την καύση του αερίου. Κυρία Πρόεδρε, μην μας περιορίζετε. Παναλαμβάνω. χρειαζόμαστε χρόνο για να μην μιλάμε μόνο για γενικότητες. Έχετε υπερβεί τα πέντε λεπτά, οπότε έπρεπε να σας διακόψω. Κυρία Χόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την ύπαρξη αυτής της έκθεσης και η κυρία Βαν Μπρέντ μίλησε για προσέγγιση no regrets η οποία με βρίσκει σύμφωνη. Μιλάμε για ανανεώσιμες και ενεργειακή απόδοση. Είναι η ραχοκοκαλιά του οδικού χάρτη για το 2050 και θα πρέπει η μελλοντική μας πολιτική να αντικατοπτρίζει αυτό το ε, δίπτυχο. Το θα πρέπει, το 2050 με συγχωρείτε, θα πρέπει να διέπεται από αυτά τα ορόσημα και θα πρέπει να τα τοποθετήσουμε στη σωστή τους θέση. Το σενάριο απανθρακοποίησης και, και τα σενάρια σε σχέση με τις μείζονες πηγές ενέργειας μιλούν για ένα 50%. Οι ανανεώσιμες αποτελούν μια ιστορία επιτυχίας το κόστος έχει μειωθεί και ο κύριος Ρόιλ μίλησε για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολλές σε αυτή τη φάση οικονομικής κρίσης. Στη Γερμανία εργάζονται πολύ περισσότεροι στις ανανεώσιμες παρά στην βιομηχανία ε, άνθρακα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία στοχοθέτηση 45% για τις ανανεώσιμες μέχρι το 2030 και έτσι η βιομηχανία μας θα μπορούσε να σταθεί πραγματικά ανταγωνιστική. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, οι ανανεώσιμες δεν θα απομακρυνθούν, αλλά θα απομακρυνθούν από την Ευρώπη. Γιατί παγκοσμίω αυξάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Μιλάμε για 40% μέχρι το 2017 παγκοσμίως, αλλά αυτή η αύξηση προέρχεται από νέες αγορές, όχι από τις ε, χώρες ε, του ΩΣΑ. Και εάν δεν δώσουμε ένα σαφές ε, μήνυμα από την Ευρώπη, τότε θα κινηθούν προς άλλες αγορές οι ανανεώσιμες και δεν θα έχουμε τις θέσεις εργασίας που επιθυμούμε. Ως προς την ε, ενεργειακή απόδοση θα θέλαμε να μειωθεί ε, το διοξίδιο του άνθρακα και η κατανάλωσή του οι εκπομπές αυτές στα κράτη-μέλη και θα θέλαμε να γίνει αναθεώρηση έγκαιρα έτσι ώστε να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι υποδομέ είναι ύψη τη σημασία θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνδεσιμότητα έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε τις ανανεώσιμες και να έχουμε μία αποδοτική, ε, ένα αποδοτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται πολλές φορές ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα backup στις ανανεώσιμες με ηλεκτροδότηση αλλά νομίζω ότι η καλύτερη βιωσιμότητα αφορά την αποθήκευση μέσω αντλιών και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης των ανανεώσιμων. Το αέριο, το φυσικό αέριο, είναι μια προσωρινή λύση βραχή πρόθεσμα. Αν μιλάμε όμως για πλήρη απανθρακοποίηση μέχρι το 2050 θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το ενδιάμεσο στάδιο, δηλαδή το 2030 και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί αυτή η τεχνολογία δεύσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα θα μπορέσει να αποδώσει μέχρι το 2030. Θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι όσον αφορά το αέριο και τις ανανεώσιμες. Θα πρέπει όμως να συνδυάσουμε το CCS με το αέριο, δηλαδή τη δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε το αέριο σαν να κλείνουμε μία βαλβίδα. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε για την μελλοντική ε, κατανάλωση φυσικού αερίου. Θα πρέπει να δούμε το αρκτικό περιβάλλον, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Θα πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε ως προς αυτό το σκέλος. Ως προς τις δαπάνες και το κόστος υπάρχει μία παρεξήγηση ότι δηλαδή οι ανανεώσιμες είναι υπέτειες για την αύξηση των τιμών αερίου. Όμως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι οι υπέτειες ε, πηγές. Μιλάμε για 300, στερλίνες αύξηση του κόστους, αλλά μόνο οι 20 στερλίνες ε, αποδίδονται πραγματικά στις ανανεώσιμες. Απλώς ε, είμαστε εξαρτημένοι δυστυχώς από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και για να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις δικές μας πηγές, ιδιαίτερα όσο αφορά τις ανανεώσιμες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τούρμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η προσπάθεια να κάνουμε έναν χάρτη πορείας ε, για την ενέργεια είναι πολύ σημαντικό, σημαντική. Γιατί? Γιατί οι ενεργειακές υποδομές έχουν κύκλο ζωής 40-45 χρόνια και επενδύσεων. Οι αποφάσει λοιπόν που θα πάρουμε σήμερα θα επηρεάσουν για παράδειγμα όσον αφορά τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα την κατάσταση του 2050. Αν φτιάξουμε τώρα ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα θα λειτουργήσει για 40-45 χρόνια. Πόσα λοιπόν, ε, πόσους ε, ηλεκτρικούς σταθμούς μπορούμε να συνδυάσουμε με CCS για να επιτύχουμε τους στόχους μας το 2050 είναι σημαντικό και για τους αγωγούς για την ηλεκτροδότηση και για την ε, μεταφορά του αερίου. Και αυτό είναι σημαντικό. Και βεβαίως, αν θέλουμε μέσω της οδηγίας για την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα να ε, μεταρρυθμίσουμε και να ε, ανακαινήσουμε και τα κτίρια μας και αυτό παίρνει, είναι μια διαδικασία που τα νέα αυτά κτίρια θα κρατήσουν 35-40 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να ξέρουμε λεπτομερώς ποια θα είναι η κατάσταση το 2050. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάποιες εξομοιώσεις. Αλλά νομίζω ότι η προσπάθεια που θα κάνουμε τώρα πρέπει να έχει ως όριο, ως ορίζοντα το 2030. Έτσι θα έχει περισσότερη έννοια. Ξέρουμε τι τεχνολογίες θα έχουμε σε όριμη φάση το 2030. Είναι η αιωλική, η ηλιακή, ήδη έχουν προχωρήσει. Μπορεί και στην ε, ε, θαλάσσια, ε, τη θάλασσα ως, τιμή, ως πηγή ενέργειας να έχουμε κάνει κάποιες σημαντικές προόδρους. Ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση επίσης και για την ανακαίνιση των κτηρίων και για τις μεταφορές ξέρουμε σε τι βαθμό θα έχουν ε, ε, αναπτυχθεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν, όταν προσπαθούμε να κάνουμε μια εξομίση το 2030, μπορούμε να την κάνουμε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Επίσης είναι σημαντικό να δούμε και τις λεπτομέρειες των προβλέψεων που κάνει η Επιτροπή. Έχουμε τρεις επιλογές No regret. Πρώτον, η ενεργειακή αποδοτικότητα πάντων θα, πάντα θα μειώνει το κόστος. Όσο πιο αποδοτική η ενέργεια, χρειάζεται και λιγότερο δίκτυο, πιο λιγότερο πυκνό δίκτυο. Περισσότερη απόδοση λοιπόν, πάντα. Καλό. Δεύτερον, και αν έχουμε πολύ CCS και πολύ πυρηνική ενέργεια, θα έχουμε πάνω από 50% ανανεώσιμες. Για την παραγωγή ενέργειας λοιπόν θα έχει μεγάλο ρόλο η αιωλική και η ηλιακή. Αυτό είναι ένα από τα κύρια μηνύματα του χάρτη πορείας. Ενώ τώρα ε, το κέντρο βάρους μας είναι συμβατικές μεγάλες εγκαταστάσεις άνθρακας πετρέλαιο, θα αλλάξει σταδιακά, δεν θα γίνει απότομα, θα αλλάξει σταδιακά προς η ηλιακή. Αυτό σημαίνει ότι η ευελιξία της αγοράς και η διασυνδεσιμότητα θα πρέπει επίσης να αυξηθούν. Σημαντικό συμπέρασμα και αυτό. Και γι' αυτό η ανακοίνωση για την εσωτερική αγορά και τον σχεδιασμό της εσωτερικής αγοράς που θα μας υποβάλει η Κομισιόν είναι πολύ σημαντική γιατί πρέπει να προκαταλάβει αυτές τις αλλαγές. Δεύτερο συμπέρασμα από την προσπάθεια εξομοίωσης. Το ανέφερε η Φιώνα. Θέλουμε περισσότερες ανανεώσιμες, περισσότερο CCS, περισσότερη, είτε πα για περισσότερη CCS, περισσότερε ανανεώσιμε ή περισσότερη πυρηνική ενέργεια, το κόστο το 2030 θα είναι περίπου το ίδιο. Δηλαδή μέσα στο ποσοστό σφάλματος είναι η διαφορά των τριών αυτών επιλογών. Αυτό σημαίνει ότι οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουμε με την πυρηνική και ο υψηλότερος κίνδυνος εκπομπών ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα που λαμβάνουμε αν πάμε για CCS δεν θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Οπότε, γιατί να μην επιλέξουμε τις ανανεώσιμες. Και αυτή είναι τώρα η πρόκληση για το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να αναλύσουμε λεπτομερώς τα στοιχεία της κάθε επιλογής ε, της εξομοίωσης και να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συνένεση για τους στόχους του 2030 και για τις πολιτικές, ε, για παράδειγμα, το σχεδιασμό της αγοράς να γίνει πιο ευέλικτη η αγορά ενέργειας, ε, παραγωγής ενέργειας. Ευχαριστώ. Ο Σιμάνσκι. Ευχαριστώ. Μία πρώτη γενική παρατήρηση. Τέτοιος στρατηγικός προγραμματισμός φυσικά έχει τεράστια πλεονεκτήματα γιατί δημιουργεί μια αίσθηση βεβαιότητας, ασφάλειας και σιγουριάς για τους επενδυτές. Αλλά θα πρέπει αυτός ο προγραμματισμός να έχει και κάποια όρια, γιατί υπάρχουν ε, προϋποθέσεις της αγοράς και τεχνολογικές που δεν μπορεί κανένα σήμερα να προβλέψει ακόμη ε, και κορυφαίοι επιστήμονες ε, και πολύ στρεχωμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να προβλέψει τους όρους ε, της αγοράς και τους τεχνολογικούς όρους του μέλλοντος. Ούτε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε και οι πιο κορυφαίοι επιστήμονες. Γιατί οι τεχνολογίες εξελίσσονται ραγδαία και μπορούν να τροποποιήσουν ρηξικέλευθα την εικόνα της ενέργειας. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε κάπως ελαστικοί και να βάλουμε κάποια όρια στο στρατηγικό προγραμματισμό. Ιδιαίτερα όταν αναφέρουμε τόσο μακροχρόνιους ορίζοντες όπως είναι το 2050. Το σχέδιο της κυρίας Τζαβέλα έχει πολλά πλεονεκτήματα, πολλές αρετές. Μ' αρέσει που ορίζει την σημασία της, των τιμών της αγοράς για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Μου αρέσει και η επισήμανση της ε, ανάγκης να λαμβάνουμε υπόψη και τα οικονομικά κριτήρια, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά την απαθρακοποίηση, την απολευθέρωση δηλαδή από το άνθρακα και την έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο και στους... εμείς ως πολιτικοί πολύ εύκολα μπορούμε να ε, μιλάμε για πολύ φιλόδοξους στόχους που μπορεί να ε, είναι λιγότερο ή περισσότερο δόκιμοι, αλλά πολλές φορές η αδύρυτη πραγματικότητα της οικονομίας μας διαψεύδει, γιατί δεν είναι δεν λειτουργεί εν κενό η ευρωπαϊκή οικονομία, λειτουργεί σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Επίσης μερικές φορές είναι ανώνυμη η οικονομία, σε τελική ανάλυση είναι οι καταναλωτές που πληρώνουν αυτό το κόστος αυτή τις ακροβασίας και ε, της διαφόρων μοντέλων που κάνουν οι πολιτικοί. Σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, σε, και σε ό,τι αφορά την αύξηση της, ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δείχνουν ότι μερικές φορές οι πολιτικές απόψεις που λαμβάνονται χωρίς, ε, οικονομική, ε, χωρίς οικονομικό υπολογισμό έχουν οδυνηρές συνέπειες όχι για τους μεγάλους παίκτες Τη ενεργειακή οικονομία, αλλά για του απλού καταναλωτέ, Γιατί ένα τέτοιο ζογκλάρισμα με τι τιμέ που γίνεται από τι πολιτικέ, μερικέ φορέ σε πολύ δύσκολη κατάσταση του απλού καταναλωτέ. Βέβαια, μερικέ φορέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ελέγξει τι πηγέ ενέργεια που θα ε, επιλέξουν τα κράτη-μέλη, αλλά επηρεάζει τη μορφή της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία της εσωτερικής αγοράς, γιατί η εσωτερική αγορά δεν μας εξασφαλίζει μόνο μεγάλη ανταγωνιστικότητα, αλλά πολλές φορές δίνει και την απάντηση, την απαραίτητη απάντηση για μια αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα πρέπει όμως να υποστηριχθεί από πιο προβλέψιμες πηγές ενέργειας και με ελαστικότητα, με ελαστικότητα, γιατί χωρίς τέτοια ελαστικότητα δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε καλά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, η διαφοροποίηση στον ενεργειακό ανεφοδιασμό είναι σημαντικό στοιχείο της ε, ε, ενεργειακής μας ασφάλειας. Δυστυχώς ε, δεν εξασφαλίζεται πάντα και στον ίδιο βαθμό τέτοιου είδους διαφοροποίηση και τέτοιου είδους ανεξαρτησία. Πολύ, σημαντικά, πολύ σημαντικές είναι οι προτεραιότητες. Ε, μερικές φορές γίνονται υπερβολικά λεπτομερικές προβλέψεις για το 2050. Επαναλαμβάνω, είναι κάπως παρακινδυνευμένο αυτό γιατί υπάρχουν αστάθμητοι και ε, απρόβλεπτοι παράγοντες και τεχνολογικοί και σε ό,τι αφορά την αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έληξαν οι σκιώδεις. και επειδή είναι τόσο σημαντικό το θέμα, υπερέβησαν όλοι τα πέντε λεπτά. Λοιπόν, ε, να ρωτήσω ποιοι άλλοι θέλουν να μιλήσουν και μετά θα κλείσω το κατάλογο μιλητών. Και πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο. Δυόμιση λεπτά λοιπόν σε αυτούς που δεν είναι σκιώδεις. Λοιπόν, ο Στάλφος Δελκαστήγιο πρώτος. Ή συνάδελφος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο που μου δώσατε. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω θερμά και να καλωσορίσω την πρόταση της κυρία Τζαβέλα, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά η πρόταση αυτή είναι ανοιχτή και μπορούμε να διευκρινίσουμε διάφορα σημεία, να προσθέσουμε νέα σημεία και είναι και ισορροπημένη ως προς το περιεχόμενό της η έκθεση αυτή. Νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι το καθήκον του εισηγητή, ιδιαίτερα σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, όπου γίνεται απλώ μια βολιδοσκόπηση ουσιαστικά των Ευρωβουλευτών. Σε ό,τι αφορά την νομοθετική δραστηριότητα για την ενέργεια στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία, είναι σημαντική, ιδιαίτερα στη δική μας Επιτροπή, γιατί η ενέργεια εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας και στα περισσότερα ντοσχέ που έχουν και νομοθετικό χαρακτήρα, ε, είδαμε ότι η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο. Τώρα έχουμε ένα ακόμη θέμα που δεν έχει νομοθετικό χαρακτήρα, αλλά έχει μεγάλη σημασία γιατί χαράζει τα βασικά στοιχεία μιας πορείας που θα είναι πολύ μακρόπνοη, έχει τεράστιο χρονικό ορίζοντα, αλλά καλό θα ήταν να πούμε από τώρα ορισμένα, σημεία, ορισμένα σχόλια για αυτό το θέμα θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για να διαμορφώσουμε το μέλλον και να χαράξουμε αυτή τη μελλοντική πορεία θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το παρόν. Δεν μπορούμε ξαφνικά να κάνουμε ένα άλμα στη μέση του δρόμου. Και ακούσαμε πριν από λίγο ότι θα πρέπει να ε, επισημάνουμε την ανάγκη ε, της ευάθυνσης στην ενιαία αγορά της ενέργειας. Αυτό είναι θεμελιώδος σημασίας όχι μόνο για λόγους οικονομικής ανταγωνιστικότητας αλλά και για λόγους ενεργειακής ασφάλειας. Και από αυτή την άποψη, το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης του ενεργειακού τομέα που εθετήθηκε το 2009 θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά και να μετατεθεί στις ε, εθνικές νομοθεσίες. Αλλιώς ε, είναι πραγματικά σαν να κάνουμε ένα άλμα στο μέλλον, χωρίς όμως ε, να ξεκινούμε και να λαμβάνουμε υπόψη το παρόν. Επιμένω λοιπόν σε αυτό. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία της παραγράφου 16, όπως πολύ σωστά κάνει η εισηγήτρια, γιατί είναι πραγματικά τεράστιος ο ρόλος του υγροποιημένου φυσικού αερίου, γιατί εξασφαλίζει τον ενεργειακό ανεφοδιασμό στην Ευρώπη. Επίσης, ήθελα να τονίσω ότι πριν αναπτύξουμε άλλους διαδρόμους, στη Μεσόγειο για παράδειγμα, θα πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν σταθμούς επανεροποίησης πολύ σημαντικούς που όμως υποτιμούνται. Αυτοί οι σταθμοί εξαέρωσης δεν αξιοποιούνται δεόντως και οι διασυνδέσεις είναι πολύ σημαντικές πριν ε, χρησιμοποιήσουμε ή κατασκευάσουμε νέες, νέους διαδρόμους. Να αξιοποιήσουμε ήδη τις εγκαταστάσεις εξαέρωσης που υπάρχουν και παραλαμβάνω υπολειτουργούν, υποχρησιμοποιούνται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μαρτσινκέβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με τον χάρτη πορείας για το 2050, αλλά θα πρέπει να βρούμε λύσεις για ε, ισότιμο καταμερισμό των δαπανών και του βάρους, γιατί ε, δεν θα θέλουμε να εκτιναχθούν στα ύψη οι τιμές ε, της ενέργειας, ε, των αδειών για την εκπορία εκπομπών. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ουδέτερη από τεχνολογική άποψη. Μέχρι τώρα πολιτικές και μέχρι τώρα λύσεις επιβαρύνουν την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα ε, ενώ υποστηρίζουν πολύ περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο προτινόμενος χάρτης για το 2050 εμβαθύνει περισσότερο στη διαδικασία αυτή και ουσιαστικά περιθεροποιεί ε, τον σημαντικό ρόλο των ορυκτών καυσίμων για την εξασφάλιση της ε, ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασμού της Ένωσης. Επίσης, σημαντικό θέμα είναι τεχνολογίες όπως το CCS, η δέσμευση αποθήκευση άθρακα, και η ενέργεια που λαμβάνεται από το όζον, που βρίσκεται σε πιλωτικό ακόμη επίπεδο. Έχουμε το Energy Outlook για το 2050 και βλέπουμε το 50% της ενέργειας στον κόσμο θα παράγεται με βάση τον άνθρακα. Και σε ό,τι αφορά το 2035 ε, θα αυξηθούν κατά 50% οι, ανάγκες, οι παγκόσμιες ανάγκες για φυσικό αέριο σε σχέση με τα επίπεδα του 2010. Οπότε μια ανεξάρτητη πολιτική μείωση της Ένωσης χωρίς ενεργειακούς εταίρους ε, από τις ε, υπόλοιπους εταίρους που χρησιμοποιούν τον άνθρακα θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Ο κοινός μας στόχος θα πρέπει να είναι η ε, ανάληψη όλων των ενεργειών προκειμένου να έχουμε αηφόρο και ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών ώστε σε, καμία ενεργεια, σε κανένα ενεργειακό τομέα να μην υστερούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Να σας ευχαριστήσω κυρία εισηγήτρια για, τη, για την παράγραφο 5 που μιλούν για την ελεύθερη χάραξη του ενεργειακού μείγματος από κάθε χώρα μέλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επίδραση που θα έχουν τα προτινόμενα σενάρια για τα κάθε κράτη, για τα, για τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι θα πρέπει στο έγγραφο αυτό να περιλάβουμε και κάποιες διατάξεις για την ε, ισότιμη αξιοποίηση των διαφόρων πηγών ενέργειας ε, και να, μεταξύ αυτών φυσικά συμπεριλαμβάνουμε και τον άνθρακα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιντάλ Κουάδρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σημαντική έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, διότι στην αρχική της πρόταση κατάφερε κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Μία γενικότερη εξισορρόπηση στόχων σε έναν τομέα όπου υφίστανται πολλά προβλήματα και διαφοροποιήσεις. Γι' αυτό αυτή η ισορροπία που μας προσφέρει στην αρχική της πρόταση ε, χρήζει επένων οι προλαλήσοντες ε, έδειξαν όλα τα σημεία μεγάλης σημασίας. Εγώ απλώς θα ήθελα να σας δώσω, να σας εκθέσω ορισμένες γενικές ιδέες ως προς τη συλλογιστική μας βάση. Όταν προγραμματίζουμε μέσο και μακροπρόθεσμα τον τομέα της ενέργειας, δεν θα πρέπει να έχουμε ιδεολογικές προκαταλήψεις. Θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, να, είμαστε, να έχουμε πρακτικό πνεύμα και να, είμα, και να μην είμαστε ιδεαλιστές. Γιατί η ιδεολογία ε, δεν αποτελεί πάντα πρόκριμα. Γι' αυτό χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η εσωτερική αγορά λοιπόν και η διάρθρωσή της είναι σημείο κλειδί για να επιλύσουμε επιμέρους προβλήματα και δεν θα πρέπει να καρκινοβατούμε τη στιγμή που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά, καθώς και ζητήματα υποδομών. Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια ε, βάση και γι' αυτό θεωρώ ότι το ενεργειακό μείγμα μας βρίσκει σύμφωνους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μία ιεράρχηση. Εάν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με το τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας ή της βιομάζας και ένα άλλο κράτος μέλος βασίζεται στα ορυκτά, τότε ο καθένας θα πρέπει να ανταποκριθεί όπως μπορεί. Να χρησιμοποιήσει κατά προτεραιότητα αυτό που ε, διαθέτει. Να μην έχουμε μια εγωιστική προσέγγιση, δηλαδή ο καθένας ορίζει το ενεργειακό του μείγμα, η κάθε χώρα ορίζει το ενεργειακό της μείγμα με βάση τις ανάγκες της. Διαφορετικά, αυτό το εγχείρημα δεν θα είχε νόημα ή θα ήταν άκρος αντιπαραγωγικό. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Ο Βιτόριο Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εργασία. Θα είμαι ιδιαίτερα συνοπτικός. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι επενδύσεις επακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Δεν πρόκειται μόνο οι τεχνολογίες, για τις τεχνολογίες που μας απασχολούν, θα πρέπει να προβούμε σε ιεραρχίες, να πούμε θα κάνουμε αυτό γιατί στοιχίζει τόσο. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ποιες είναι οι εμπλεκόμενες επενδύσεις για κάθε σχήμα και να μιλήσουμε για τρόπους εφαρμογής των επενδύσεων. Αυτό, αυτό το πνεύμα θα πρέπει να μας διέπει. Να μιλάμε δηλαδή για χρηματοδοτήσεις τύπου ευρωομολόγων ή ομολόγων έργου. Γιατί οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν γιατί έτσι θα υπερβούμε αυτή την δύσκολη φάση οικονομικής ε, κρίσης που διανύουμε. Μιλάμε για τεχνολογικά μέσα, θα πρέπει όμως να κάνουμε μία πρόβλεψη για το μέλλον, γιατί δεν μπορούμε να επενδύσουμε στον άνθρακα τη στιγμή που το εμπλεκόμενο κόστος είναι πολύ υψηλό και αυτό αφορά και το CCS, την αποθήκευση, τη δέσμευση και την αποθήκευση, γιατί ε, αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της ε, πίτας και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε από πλευράς επενδύσεων. Αυτό αφορά και το ETS, δηλαδή την ε, ανταλλαγή εκπομπών αερίου. Και χτες μιλήσαμε και για ένα παράπλευρο ζήτημα, δηλαδή τα ενεργειακά δίκτυα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε φαρετά την κατάσταση γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης και έτσι θα μειώσουμε την αποθήκευση ενέργειας ενώ θα βελτιστοποιήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ως προς τις, ε, το σχήμα εμπορίας, ανταλλαγών δηλαδή, το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS, σας δείχνω μία δημοσίευση του ε, Policy Department όπου έχει τίτλο Much Ado About Nothing, πολύ θόρυβος για το τίποτα σε σχέση με το ε, Ρίο Συνήκωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως προς τις εκπομπές και υπάρχει και σωρία άλλων στοιχείων που θα πρέπει να μας απασχολήσουν Ήδη πολλά ελέγχθησαν από τους προλαλήσαντες και εγώ θα υποβάλω συγκεκριμένες τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Χίμπνερ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έγγραφο που θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις στον ενεργειακό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Τζαβέλα, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό το έγγραφό της και ε, χαίρομαι που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ελαστικότητα, γιατί χρειάζεται ελαστικότητα για να δημιουργεί κάθε χώρα το δικό της ενεργειακό μείγμα. Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι είναι και σημαντικό για την Ευρώπη, δηλαδή τη μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε γενικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, χαίρομαι που ελήφθησαν υπόψη κάποια σημεία προκειμένου να διασκεδαστούν ε, κάποιες ανησυχίες μας, γιατί μερικοί φοβόμασταν ότι ορισμένες χώρες θα περιθωριοποιηθούν και θα αφηθεί καθεμία στη μοίρα της για να αντιμετωπίσει τα ενεργειακά της προβλήματα. Ιδιαίτερα οι χώρες που χρησιμοποιούν τον λιθάνθρακα ή τον γιάνθρακα ως βασικό στοιχείο του ενεργειακού τους μείγματος. Είναι πολύ σημαντικές τεχνολογίες όπως η τον γιανθρακα ως βασικο στοιχειο του ενεργειακου του μειγματος ειναι πολυ σημαντικες τεχνολογιες οπως η δεσμευση και η αποθήκευση του άνθρακα και άλλες τεχνολογίες που αφορούν ε, ορυκτούς πόρους, γιατί και αυτές οι τεχνολογίες μας δίνουν την ε, δυνατότητα να απτυχθούμε σε ενεργειακό επίπεδο. Από αυτή την άποψη ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια για την ελαστικότητά της. Μην ξεχνάμε αυτά που είπαμε χθε για το COP18 και οι συνάδελφοι εξέφρασαν κάποιε ανησυχίε μπορούμε να μειώσουμε το κόστο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εισάγοντας για παράδειγμα ηλιακού θερμοσορευτές από την Κίνα. Αλλά δεν είναι λύση αυτή, γιατί έτσι θα έχουμε εξαγόμενε εκπομπέ. Γιατί οι ηλιοθερμοσορευτέ τη ε, Κίνα και τα ηλιακά πάνελ που παράγονται στην Κίνα δεν τηρούν τι ίδιε υψηλέ περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ με εμά. Δεν θα πρέπει έτσι να οδηγήσουμε σε μετεγκατάσταση των δικών μας βιομηχανιών και ταυτόχρονα να εισάγουμε ε, προϊόντα που ε, ε, εκπέμπουν πολύ περισσότερα καυσαέρια. Προσοχή λοιπόν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θα πρέπει να μετακυληθεί το κόστος τους σε άλλα σημεία και ιδιαίτερα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη ενεργειακού, ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασμού στην Ευρώπη. Και προ, ε, ε, θέλουμε παρακαλώ να μην στερήσουμε από τους δικούς μας παραγωγούς την, ενέργεια, την δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζόρνταν έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν μιλάμε για έγγραφα της Επιτροπής, όταν συζητάμε έγγραφα της Επιτροπής, πολύ συχνά λέμε ότι είναι καλή βάση και μετά προσθέτουμε και άλλους στόχους στα κείμενα αυτά και τα αλλάζουμε όλα. Σε αυτή την περίπτωση όμως καλύτερα να εξετάσουμε προσεκτικά τις ανάγκες μας. Γιατί πρέπει να κάνουμε συμπληρωματικούς υπολογισμούς. Πρέπει να καταλάβουμε τι κόστος θα υπάρχει σε κάθε σενάριο, για παράδειγμα, εάν δεν υπάρξει διεθνής αλλαγή, παγκόσμια αλλαγή για την παγκόσμια δράση για την κλιματική αλλαγή, τότε δεν θα είναι εύκολο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει μόνη της. Εάν ε, συνεργαζόμασταν με άλλους θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική η δράση μας. Πρέπει λοιπόν να μας δώσει συντοματική πληροφόρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ρόιλ προηγουμένως. Πρέπει ε, να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι. Να καθορίσουμε τους στόχους μας και μετά να τους μελετήσουμε. Είμαι η συγγήτρια της Επιτροπής ΕΝΒΗ και προτείνω ένα μόνο στόχο, στόχο για το διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά να δούμε τι άλλους στόχους χρειαζόμαστε για να μειώσουμε τις εισαγωγές που κάνουμε στον ενεργειακό τομέα. Δεν χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη στον ενεργειακό τομέα, περισσότερη, αλλά βασιζόμενοι στους μηχανισμούς της αγοράς. Και κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Οποιασδήποτε επιδοτήσεις πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένες. Κάποιες επιδοτήσεις θα πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικές κάποια στιγμή. Να μπορούν τα, να σταθούν μόνες τους στα πόδια τους. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να τις επιδοτούμε επαόριστον. Επίσης, για να καθορίσουμε τους στόχους μας, να καταλάβουμε τις ιδιαιτερότητες των μικρών συστημάτων ενέργειας. Εάν περιορίσουμε τη δυνατότητα χρήση αυτών των στόχων, στην ουσία ε, θα είναι πολύ άκαμπτη η χρήση των μικρών συστημάτων ενέργειας. Διότι ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ε, μεγάλη κλίμακα συστήματα είναι πολύ διαφορετικό από τα μικρή. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, η αλληλεπίδραση των διαφόρων ενεργειακών πολιτικών και των διαφόρων κρατών μελών είναι πρωταρχική σημασία. Θα πρέπει να μα βοηθήσει και η υπηρεσία ACER για τη συνεργασία των ρυθμιστών στον τομέα αυτό. Απαραίτητο επίση, είναι καλύτερη συμπερίληψη των μεταφορών και τη θέρμανση σε αυτόν τον χάρτη πορείας και επίσης ο ορίζον 2020. Ελπίζω η ενέργεια να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο αυτό του 2020 και πρέπει να είμαστε όσο ουδέτεροι όσο γίνεται. Ευχαριστώ. Κορέγια του Κάμπος. Πέντε ιδέες θα ήθελα να εκθέσω. Καταρχήν, αυτό το εγχείρημα του οδικού χάρτη είναι πολύ σημαντικό. Μας βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνος και νομίζω ότι η έκθεση Τζαβέλα στέκεται στα πιο σημαντικά σημεία. Τώρα, υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία τα οποία δεν είναι μετρήσιμα Καταρχήν ως προς τα πυρηνικά, βλέπουμε ότι κλείνουν στην Ιαπωνία. Δεν ξέρουμε αν θα ξαναανοίξει η μονάδα της ε, Φουκουσίμα και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι τιμές θα αυξηθούν και παράλληλα υπάρχουν και στοιχεία που μας δείχνουν ότι το κόστος του φυσικού αερίου επιμερίζεται στο 5. Επίσης, οι ΕΠΑ προβάλλουν τη δική τους πολιτική και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε. Όλη αυτή η ενεργειακή πολιτική έχει επιπτώσεις και στη βιομηχανία. Τα ευρωπαϊκά δηληστήρια δεν σχετίζονται, δεν αλληλοσυνδέονται με επιχειρήσεις διανομής και κλείνουν το ένα μετά το άλλο, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος και επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Έχω πολλές αμφιβολίες για το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στην Ευρώπη. Η κυρία ε, Τζαβέλα αναφέρεται στα δηληστήρια στην έκθεσή της και νομίζω ότι θα πρέπει να επεκταθούμε. Τώρα, ως προς την εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών, αυτό είναι ε, το τέταρτο στοιχείο. Πρόκειται για έναν τέταρτο αστάθμητο ε, παράγοντα για το κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε το κόστος. Ξεχνάμε τα δικαιώματα των καταναλωτών πολύ συχνά. Φαίνεται ότι το ενεργειακό μείγμα και η ενέργεια αποτελεί μία μορφή φορολογικής μόλυνσης και δεν υπάρχει επαρκής οικονομική ανάλυση. Υπάρχουν ορισμένα προβλέψιμα στοιχεία και γνωρίζουμε πώς έχει η ζήτηση, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η προσφορά. Σας ευχαριστώ. Σκίνερ. Μα δεν ζήτησα το λόγο. Ευχαριστώ που μου το δίνετε παρόλα αυτά. Εκπλήσω με λίγο. Υπερβάλλον ζήλος από τη δική μου πλευρά. Ο κύριος Ζαντό, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Μια παράθεση θα θέλω να κάνω. Του Μπαράκ Ομπάμα το 2009 είπε «Έχουμε λοιπόν επιλογή. Μπορούμε να μείνουμε η πρώτη εισαγωγή ε, πετρελαίου στον κόσμο και να στέλνουμε τα λεφτά μας και το πλούτο μας στο εξωτερικό ή να γίνουμε η πρώτη εξαγωγή ε, καθαρής ενέργειας. Μπορούμε να αφήσουμε τους ανταγωνιστές μας να πάρουν τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος ή μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της εποχής μας. Η χώρα που θα είναι ηγετική στις καθαρές τεχνολογίες θα είναι η χώρα που θα ηγείται της διεθνούς οικονομίας τον 21ο αιώνα. Μέχρι στιγμής η Ευρώπη είχε επιχειρήσει να είναι και στα δύο, να είναι ανάμεσα σε δύο καρέκλες. Και φιλόδοξοι στόχοι για τις ανανεώσιμες μπορούμε να κάνουμε όλο και περισσότερα και μια, ένας κλάδος ε, βιομηχανικός των ανανεώσιμων που είναι ε, αρκετά καινοτόμο. Δηλαδή, αντίθετα, ε, είχε προχωρήσει ε, διτά στο σωστό δρόμο. Τώρα πάμε όμως πίσω σε παλιέ ενέργειες και συμβατικές όπως και στο λιθικό φυσικό αέριο και μειώνεται η ανταγωνιστικότητά μα στις ανανεώσιμες όπου υπάρχει έντονη ανταγωνιστικότητα κυρίως από την Κίνα. Να μην επιλέξουμε λάθος σύγκρουση. Εάν πληρώνει τόσο ακριβά η Ιαπωνία σήμερα την ενέργειά τη, είναι επειδή στράφηκε αποκλειστικά και τυφλά προς ε, την πυρηνική ενέργεια. Κάθε χρόνο δαπανούμε 188 δισεκατομμύρια για ενέργεια που εισάγουμε από το εξωτερικό, ενώ οι ανανεώσιμες είναι καλές και για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για την απασχόληση. Ένα τελευταίο στοιχείο. 488 εκατομμύρια, 488 εκατομμύρια για εισαγωγές εάν το μέσο κόστος μια θέση εργασίας είναι 30.000 ευρώ, είναι 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 15 εκατομμύρια χάνονται επειδή δεν δρούμε αρκετά για ε, οικονομίες στην ενέργεια και για ανανεώσιμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που απουσίασα από την ψηφοφορία, αλλά είχα ψηφοφορία σε μια άλλη επιτροπή. Είναι πολύ δύσκολο έργο να θεσπίσουμε ένα στόχο που θα υλοποιήσουμε μετά από 40-50 χρόνια χωρίς να ξέρουμε με τι θα είναι σπαρμένη αυτή η πορεία, γιατί υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες και πολλές αβεβαιότητες. Και αυτό είναι το δυνατό σημείο της έκθεσης. Το άνοιγμα, η ελαστικότητα προς διαφορετικές μορφές ενέργειας και διαφορετικές εφευρέσεις και έρευνες. Γιατί θα πρέπει να αφιερώσουμε πολύ μεγαλύτερο τμήμα του προπολογισμού μας και για την καινοτομία και για την τεχνολογία, αλλά και για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και φυσικά στη συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλές καινοτομίες στον τομέα της ενέργειας. Επίσης θα αφιερωθούν πολύ περισσότερα κονδύλια σε ενεργειακά προγράμματα από ό,τι σήμερα. Να μην λέμε από τώρα δηλαδή ποιο θα είναι το ενεργειακό μέσων του μέλλοντος. Γιατί μιλάμε για το μέλλον κύριε Ζαντό, δεν μιλάμε για το παρελθόν. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι μελλοντικέ ενεργειακές πηγές. Απλώς ε, ε, μπορούμε να εικάζουμε, να συζητούμε, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα. Ας αφήσουμε λοιπόν ελεύθερο το πεδίο, να μπορούμε να δημιουργήσουμε συνεργασία και συνδυασμό των διαφορετικών πηγών ενέργειας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι σημαντικό να συμπληρωθεί αυτό το ε, χάρτης πορεία με τους εθνικούς χάρτες πορεία. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο ένα χάρτη πορεία, κομμένο και ραμμένο, one size μάλλον που θα ταιριάζει σε όλους. Χρειαζόμαστε και ε, τους εθνικούς χάρτες πορείας. Υπάρχει μια απόπειρα ε, τέτοιων χαρτών πορείας ε, με χαμηλή χρήση άνθρακα. Αυτό όμω είναι άλλο θέμα, ένα άλλο έγγραφο και θα πρέπει ίσως να το λάβουμε υπόψη στη συζήτηση και να το συνδυάσουμε. Δεν θέλω να μακρηγορώ. Έρχομαι στο τελευταίο μου σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημιούργησε μια, ένα peer review, μια ε, ε, ε, αξιολόγηση από ισότιμους. Υπάρχει αυτό το έγγραφο, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν δεόντως τα πορίσματα αυτού του peer review. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επισυναυθούν στην έκθεση αυτά τα πορίσματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά και καλό θα ήταν να ληφθούν υπόψη και στο δικό μας χάρτη πορείας. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία εισηγήτρια, κυρία Τζαβέλα, τους Σκιώδης ε, και τους άλλους που πήραν το λόγο. Για μας ε, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να ακούσουμε τη συζήτηση και φυσικά και η έκθεση. Ο χάρτης πορείας 2050 δεν ασχολείται τόσο πολύ με το τι θα γίνει το 2050, αλλά το πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Όπως ξέρετε, οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα είναι μακροπρόθεσμες, οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σήμερα και γι' αυτό αναλύσαμε με τη βοήθεια διαφόρων εναλλακτικών λύσεων τι πρέπει να γίνει. Η κατάσταση στα κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετική, το μείγμα είναι θέμα κάθε κράτος μέλος, αλλά παρόλα αυτά με τη βοήθεια των εναλλακτικών καταλήξαμε σε αυτές τις λύσεις no regret, όχι μετάνοια, που τις καλωσορίσανε διάφοροι. Χρειαζόμαστε ανανεώσιμες, χρειαζόμαστε αποδοτικότητα, αλλά χρειαζόμαστε και υποδομές και εσωτερική αγορά. Γι' αυτό η Κομισιόν θα κάνει με βάση τον ε, χάρτη πορεία τρεις ανακοινώσεις. Μία έχει ήδη γίνει για τις ανανεώσιμες, η δεύτερη το φθινόπωρο για την εσωτερική αγορά που θα γίνει και ανάλυση και ανακράτος μέλος και θα υπάρξει μία τέλη αρχές του επόμενου για την σημασία του CCS, αποθήκευση, ε, δέσμευση, ε, αποθήκευση. Όσο πιο συγκεκριμένη η έκθεση στα συγκεκριμένα αυτά θέματα, τόσο καλύτερη για μας, γιατί το επόμενο βήμα που θα είναι το 2013 ε, είναι το 2030. Είμαστε ανοιχτοί για το κείμενό μας για το 2030. Χρειαζόμαστε περαιτέρω φυσικά αναλύσεις, τι στόχους θα επιλέξουμε το 2030 και τι είναι αναγκαίο. Αλλά σήμερα συζητάμε για τον χάρτη 2050 Φυσικά όσα είπατε θα λάβουμε υπόψη, είναι σημαντικά και καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει και μια κρόαση όπου φυσικά θα συμμετάσχει ενεργά η Κομισιόν και ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η εισηγήτρια, η κυρία Τζαβέλα, για να συνοψίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρος και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις επικοδομητικές ε, προτάσεις τις οποίες κάνανε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάτι. Ε, καλούμαστε να συντάξουμε μία έκθεση στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Η Επιτροπή είναι βιομηχανία, ενέργεια και ε, research and development. Ε, σας ομολογώ προσωπικά ότι αν ήμουνα ένας επενδυτής στην ενέργεια ή στη βιομηχανία ή στην έρευνα στην Ευρώπη και διάβαζα το κείμενο το οποίο σας έχω υποβάλει, δεν θα ήμουν σίγουρος αν, που και αν θα έπρεπε να επενδύσω. Είχα μεγάλη δυσκολία να βάλω σε μία ρεαλιστική βάση το κείμενο και να δώσουμε συγκεκριμένες, να δώσω μέσα από αυτό το κείμενο συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τους επενδυτές, τους Ευρωπαίους επενδυτές στη βιομηχανία και στην ενέργεια. Για το λόγο αυτό σας έχω διανύμει συνημένα μία λίστα με γιατί είχα και το, τον περιορισμό των ε, λέξεων μία λίστα με που ίσως βοηθήσουν να γίνει το κείμενο καλύτερο. Αλλά βασίζομαι και στη δική σας στήριξη και σε αυτά τα οποία θα προτείνετε να διαμορφώσουμε το κείμενο για να κάνουμε ένα κείμενο όμως ρεαλιστικό και το οποίο πράγματι θα δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι πρέπει να γίνει στην ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της ενέργειας, αλλά να είμαστε συγκεκριμένοι. Μιλήσατε για ελαστικότητα, δεν επέδειξα ελαστικότητα, ήθελα να είμαι ρεαλίστρια. Θέτω ένα ερώτημα. Αν δεν υπάρξει παγκόσμια δράση για το κλίμα, τι πρέπει να κάνουμε. Το θέτω ως ερώτημα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να συζητήσω είναι να υιοθετήσουμε όλοι ότι μέσα από αυτό το κείμενο θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το μεταβατικό στάδιο αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν με στόχο το 2030 και για το 2050. Θα έχουμε λοιπόν ένα μεταβατικό στάδιο με τους στόχους που έχουμε θέσει για τις ανανεώσιμες μέχρι το 50. Πρέπει να λάβετε υπόψη όλοι ότι δεν μπορεί να αγνοήσουμε το ρόλο τον οποίο παίζουν διάφορα άλλα προϊόντα στην ενέργεια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο που θέλουμε το 2050. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το αέριο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αν υπάρχουν δικές μας ευρωπαϊκές πηγές ενέργειας. Θα μιλήσουμε και για το shale gas, θα έχουμε και την αναφορά. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αν υπάρχουν καινούρια μέρη όπου μπορούμε να αντλήσουμε αέριο ή ακόμα και πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο δεν θα εξαφανιστεί μαγείας. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θέλω επίσης να επισημάνω το εξής. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του οικονομικού ή και πολιτισμικού θα έλεγα επίπεδου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει κάποιες χώρες να καταλάβουν ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν μεγάλες ανάγκες, είναι πολιτισμικά, θα έλεγα λίγο πιο πίσω, και θα πρέπει να εκπαιδευτούν και στο θέμα του περιβάλλοντος. Γι' αυτό βάζω ότι θα πρέπει να βάλουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα στη δημόσια εκπαίδευση και θα πρέπει να δείξουμε μία κατανόηση ότι είμαστε 27 κράτη-μέλη και τα οποία θα κινηθούμε στο 2050 με διαφορετική ταχύτητα επιτυχίας και επίτευξης στόχων. Οφείλουμε λοιπόν να κινηθούμε πιστεύω μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να ξεκαθαρίσουμε πράγματι την ενεργειακή μας πολιτική η οποία, η οποία παίζει τεράστιο ρόλο στην διαβίωση ή ακόμα και στην επιβίωση του Ευρωπαίου πολίτη. Κάποια κράτη-μέλη έχουν πολυτέλειες να υιοθετήσουν κάποιες άλλες ενεργειακές συμπεριφορές. Κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν την έχουν αυτή την πολυτέλεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να ζητήσω την βοήθειά σας να κάνουμε ένα όσο μπορούμε πιο ξεκάθαρο κείμενο για το 2050 θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση των στόχων του 2020 για να βοηθηθεί και να είναι ρεαλιστικό το 2030 που θα βγει από την Επιτροπή και μέχρι ότου διαμορφώσουμε το κείμενό μας θα έχουμε αρκετά στοιχεία ούτω ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο πραγματικοί και ρεαλιστές σε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Τζαβέλα. Η ακρόαση αποφασίστηκε από τους συντονιστές για τις 18 Σεπτεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 5 και οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Okay, the... Το επόμενο θέμα είναι ο Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπουτικόφερ, τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Γερμανός Αν δεν σε ενδιαφέρει ο προπολογισμό. Μάλλον κάνετε λάθο. Έχω εμπλακεί εδώ και δύο χρόνια με τις διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή Προπολογισμών αλλά ποτέ δεν ε, ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση όσο τώρα και θα σας καλούσα Πρόεδρο. παρακαλώ κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να αποχωρήσετε, παρακαλώ ε, να εξέλθετε. Κύριε Μπιτικόφερ. Δεν ακούγεται. Θα σας καλούσα να να ακούσετε αυτά που έχω να σας πω για την κατάσταση που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ιδιαίτερα δύσκολη η εξέβρεση λύσης. Η Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού που ενέκρινε τον Απρίλιο προέβλεψε μια συνολική αύξηση 2% στις δεσμεύσεις, στις υποχρεώσεις, δηλαδή το επίπεδο του πληθωρισμού και αύξηση 6,8% στις πληρωμές για να σεβαστεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της, του τρέχοντος και παρελθόντων ετών. Για την ε, κατηγορία 1α, για τον τίτλο 1α, ανάπτυξη και απασχόληση, η αύξηση υποχρεώσεων υποτίθεται πως έπρεπε να είναι 4,1% και η αύξηση των, των πληρωμών 17,8%. κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στο ότι έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές μας, τις συμβατικές υποχρεώσεις των κληρονών μας. Για το ΣΥΠ, ανταγωνιστικότητα και ε, καινοτομία γύρω στο 7% ήταν η αύξηση. Χαμηλότερο δηλαδή από ότι ήταν η νομική βάση και το, πρόγραμμα, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Μετά την ε, έκφραση άποψη από το Κορεπέρ, το σχέδιο προπολισμού του Συμβουλίου στον τίτλο 1α αντί για συν 4 στις υποχρεώσεις θα είναι μόνο συν 1,5% και αντί για συν 17 στις πληρωμές μόνον συν 1,04. Δηλαδή, κατά την άποψη του Συμβουλίου, οι αυξήσει θα είναι περίπου στο ίμιση του πληθωρισμού. Η περικοπή των πληρωμών εντός του ε, προγράμματος SIT του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας θα είναι πολύ μεγάλη. Αυτό είναι απόλυτα αντίθετο με τους στόχους του Συμφώνου για Ανάπτυξη και Εργασία που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών πολύ πρόσφατα. Είπαν ότι πρέπει να ενισχυθεί η ενίσχυση της έρευνας ανάπτυξης των δυνατοτήτων επένδυσης. Είπαν ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα startup που έχουν καινοτομίες και τώρα μας δίνουν ένα προπολογισμό που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις εκκλήσεις τους οι περικοπές του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και κοινοτομίας, εάν γίνουν, θα οδηγήσουν σε ιδιαίτερη επιδείνωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων στις επενδύσεις, τώρα που τη χρειάζονται. Και η περικοπή στις πληρωμές θα οδηγούσε στην ε, διακοπή του προγράμματος, της εφαρμογής του προγράμματος. Όπως είπε η Επιτροπή, οι τιμές για τις, ε, τα ποσά για τις υποχρεώσεις προβλέπει το Συμβούλιο θα είχαν λήξει τον προσεχή Μάιο. Στην έκθεση Λαβία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο ως βάση για τον τριμερή διάλογο όλοι ψηφίσαμε υπέρ ισχυρής υποστήριξης ενός επαρκούς επίπεδου ε, πόρων στον ε, προπολογισμό του 2013 υπέρ ε, υπεύθυνης ε, ε, συμπεριφοράς και κατά τεχνητών περικοπών και ιδιαίτερα υπέρ της λήψη υπόψη των πραγματικών αναγκών και πόρων για να φτάσουμε στους διακηρυγμένους στόχους μας και υπέρ της υποστήριξης, της ανάπτυξης και τη ε, απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους και τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το 2013. Κανείς από αυτούς τους στόχου δεν μπορεί να επιτευχθεί με, το στόχο όπως, με τον προϋπολογισμό όπως τον αποφάσισε το Συμβούλιο. Σαφεί λοιπόν οι εναλλακτικέ λύσει. Ή σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και καθιστάμεθα συνυπεύθυνοι για το ότι οι μικρομεσαίες και η ανταγωνιστικότητα θα καταρακωθούν σε συνθήκες κρίσης ή, ή οπλιζόμεθα για έντονη σύγκρουση με το Συμβούλιο. Βέβαια, τη μάχη δεν θα την κάνω μόνο εγώ ή μόνο η Επιτροπή μας. Ή, ή την επιλογή καλύτερα. Αλλά δεν με ενθαρρύνει ιδιαίτερα το ότι ελάχιστοι θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουν καν αυτά τα οποία λέω όταν συζητιούνται τα θέματα αυτά στην ημερήσια διάταξη. Κοιτάξτε, δεν θα τα βάλω με όλους. Βλέπω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και μπορώ να παραπονεθώ και θα είχα εγώ ε, μικροπολιτικό όφελος. Αντίθετα θα προτιμούσα να συστρατευτούμε για να επιχειρήσουμε να αποφύγουμε τις ε, ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις των προτάσεων του Συμβουλίου. Ενημέρωσα τους κοιόδης τις αλλαγές που θα πρότεινα στον προϋπολογισμό. Δεν θέλω να αποκαταστήσω όλη την ε, αρχική πρόταση της Κομισιόν, θα μπορούσα να υποχωρήσω σωσμένα στοιχεία, αλλά προσπάθησα να αποκαταστήσω όλες τις θέσεις του προπολογισμού που αφορούν έρευνα ανάπτυξη, μικρομεσαίες και αυτή θα πρέπει να είναι η κόκκινη γραμμή για μας, για την Επιτροπή μας. Αυτό θα ήθελα, τουλάχιστον εγώ να προτείνω. Η εργασία μας για την ε, αντιμετώπιση του προπολογισμού θα είναι δυσχερής. Θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 3 Σεπτεμβρίου. Άρα δεν υπάρχει χρόνος γιατί έχουμε διακοπές ενώπιών μας για συνάντηση των σκιωδών. Οι συνάδελφοι καλούνται να υποβάλουν τροπολογίες ε, προθεσμία 21 Αυγούστου. Κάτι ακόμη για τα πιλωτικά προγράμματα. Υπάρχουν 7 πιλωτικά προγράμματα. Έχουν προταθεί από μέλη της Επιτροπής μας 7 πιλωτικά προγράμματα. Τρία εκ των οποίων έλαβαν βαθμό Α κατά την αποτίμηση της Επιτροπής. Θα πρότεινα λοιπόν η Επιτροπή μας εν ευθέτω χρόνο να ψηφίσει πέρα αυτών των τριών προγραμμάτων που πήραν τον καλύτερο βαθμό. Τα υπόλοιπα προγράμματα πήραν C και D βαθμό, οπότε προτείνω να τα καταλήψουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μπιτικόφερ. Δεν έχουμε κανένα σκιώδη εκπρόσωπο ούτε από το ΕΛΚ ούτε από τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, δεν ξέρω αν ο κύριος Σκίνερ θέλει το λόγο. Νομίζω ότι ο κύριος ε, Μπουτικόφερ μας έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα σκιαγράφηση ε, της κατάστασης και συμμερίζομαι τις ανησυχίες του, ιδιαίτερα για το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, Ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Χρειαζόμαστε επενδύσει, ε, βρισκόμαστε σε ένα ζωφερό οικονομικό κλίμα και ε, διαρωτώ με κατά πόσο η Επιτροπή Προϋπολογισμών αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης περιορίζοντας τις καινοτομίες και τις επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Νομίζω ότι εμείς είμαστε πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα, γι' αυτό ενθαρρύνω τον κύριο Μπουτικόφερ να συνεχίσει την προσπάθειά του παρά την φανή έλλειψη ενδιαφέροντος από τους συναδέλφους. Βέβαια, δεν εκπροσωπούνται εδώ πολλές ομάδες. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αποθαρρύνεστε κύριε Μπουτικόφερ. νομίζω ότι και η Επιτροπή Προπολογισμών δείχνει βέβαια ρεαλισμό συνήθω, αλλά θα πρέπει να έχει υπόψη ότι υπάρχουν ανάγκες για περισσότερες επενδύσεις για ορισμένε επιτροπέ. Θα πρέπει επιτέλους, για να ξεφύγουμε από την κρίση, μερικές φορές να ξοδέψουμε και περισσότερα και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συνεχίσει τις πιέσεις για να επανέλθουμε σε πιο ε, σημαντικές επενδύσεις και πιστώσεις γιατί ελπίζω οι οικονομίες να είναι διοικητικές και όχι σε περικοπές ε, σε σχέδια, γιατί περικοπές σε σχέδια ισοδυναμούν με λιτότητα και όχι σε επενδύσει στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης και την καινοτομία. Ευχαριστώ κύριε Σκίνερ. Ε, θα, θα πάρω εγώ ίδιο το λόγο γιατί είμαι σκιώδης ηγητής της Άλντε. Η Άλντε έχει ξεκάθαρους προσανατολισμούς και προτεραιότητες στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Καταρχήν, η δημοσιονομική ε, σοφία και προφυλακτικότητα που έδειξαν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχει ένα αντίκτυπο και να αντικατοπτρίζεται και στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Γιατί είναι προκλητικό να συρρυκνώνουμε και να περικόπτουμε αδρά τους εθνικούς προϋπολογισμούς και να επιτρέπουμε αύξηση γύρω στο 7% στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Βέβαια δεν υπάρχουν ιερές αγελάδες όταν χρειαζόμαστε ε, δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά θα πρέπει να είμαστε ευφύς στον τρόπο που επιβάλλουμε τις περικοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πολιτικές προτεραιότητες, υπάρχει ευρεία συνένεση ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η καινοτομία και η έρευνα είναι το κλειδί για την οικονομική μας ανάπτυξη. Είμαστε υπέρ ε, τη αύξηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για, τα, ε, για το, πρόγραμμα, το πρόγραμμα πλαίσιο και το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση σε όλε τι δημοσιονομικέ γραμμέ. Εμεί δεν είμαστε υπέρ γενική αύξηση του κοινοτικού προπολογισμού, αλλά για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη είμαστε υπέρ τη αύξηση των κονδύλιων. Τώρα, πώς θα δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια. Βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε προς το επόμενο ε, να ε, χρηματοδοτήσουμε περισσότερα ε, προγράμματα επίδειξης και επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια για μόχλευση και για προσέλκυση και των ιδιωτικών κονδύλιων. Έχουμε πιλωτικά προγράμματα στο 2013 για ομόλογα έργο, Πολύ σωστό, γιατί θα συνεχιστούν οι επενδύσεις στο μέλλον μας ουσιαστικά, ενώ ταυτόχρονα ε, θα προσπαθήσουμε με λιτότητα των προπολογισμών και λαμβάνοντας υπόψη και την προοπτική της αγοράς να χαράξουμε τις κοινοτικέ πολιτικές. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχει κανείς. Ο κ. Μπουτικόφερ έχει το λόγο για να συνοψίσει. Δεν είναι σημαντικό το θέμα. Τι να συνοψίσω. Okay. Well, still we uh, need to vote. Πρέπει να ψηφίσουμε στις 3 ε, Σεπτεμβρίου. Προβλέπεται η ψηφοφορία και η υποβολή τροπολογιών ε, είναι μέχρι τις 21 Αυγούστου, όπως είπε ο κύριος Μπουτικόφερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε Προεδρία. Bene. Inizia... Ringraziamo... Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταύρο Μαλά, Υπουργό Υγείας, αρμόδιο για το χαρτοφυλάκιο της έρευνας και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται μεταξύ μας σήμερα βρίσκεται μαζί μας σήμερα για να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Έχουμε 45 λεπτά για τη συζήτηση και για να γνωρίσουμε τις προθέσεις της νέας Προεδρίας και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να υποβάλουμε ερωτήσεις προς τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, έχετε στη διάθεσή σας 10 με 15 λεπτά και μετά θα σας υποβληθούν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προτιμούσα να είχα περισσότερο χρόνο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον συζήτηση που κάνουμε για την έρευνα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, νιώθω, οπωσδήποτε ιδιαίτερη χαρά για την ευκαιρία που μου δίνεται να παρουσιάσω ενώπιον της Επιτροπής σας σήμερα για να παρουσιάσω το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας της Κύπρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Συζητώντας αυτό το θέμα, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι η δήλωση της Αβώνας το 2001. Τότε είπαμε στους πολίτες της Ευρώπης ότι μέχρι το 2010 η Ευρώπη θα γίνει η πιο δυναμική οικονομία στον πλανήτη με την έρευνα και την καινοτομία να είναι στην καρδιά αυτής της έρευνας. 11 χρόνια αργότερα έχουμε μια έντονη οικονομική κρίση που κάνει τα θεμέλια πολλών κοινωνιών να τρίζουν με διάφορους τρόπους. Η νέα, η στρατηγική για το 2020 θεωρεί ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι από τις βασικές, ε, βασικούς τομείς της δραστηριότητάς μας. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε σωστά και απτά πολιτικά μηνύματα στους πολίτες μας. Αναμφίβολα, η διέξοδος από την κρίση είναι μέσα από την ανάπτυξη, τις πολιτικές που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο που συμπίπτει με τις διαπραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα ενέργειας για την έρευνα και την καινοτομία που είναι γνωστός ορίζον 2020. Έχουμε συνέστηση των καθηκόντων μας και προσβλέπουμε σε επικοδομητική συζήτηση και στο Συμβούλιο αλλά και ακόμη πιο σημαντικό προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως αναμένεται, ο ορίζον 2020 είναι αναμφίβολα η πρώτη μας προτεραιότητα. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, θα ασχοληθούμε και με τρία άλλα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ε, Καινοτομία και την Τεχνολογία, EIT, που είναι τμήμα του ορίζοντα 2020, του νομοθετικού πακέτου, τον Ευρωπαϊκό ε, Χώρο Έρευνας, ERA, και τη διεθνή συνεργασία για την έρευνα και την καινοτομία με ιδιαίτερη εστίαση στην ευρωμεσογειακή διάσταση. Για τον ορίζοντα 2020 και το νομοθετικό του τμήμα, το Συμβούλιο ε, ακολουθεί μια προσέγγιση κατά τμήματα ε, ε, για την εξέταση των προτάσεων, ενώ το Κοινοβούλιο προτιμά να τα εξετάσει ως δέσμη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την ε, Δανέζικη Προεδρία που ε, κατέληξε σε συνένεση στο Συμβούλιο για το πρόγραμμα για την ε, δομή και τα σημεία κλειδιά, δηλαδή για το κύριο πρόγραμμα πλαίσιο και τον κανονισμό για αυτό τον περασμένο Μάιο. Η συμφωνία το Μάιο στο Συμβούλιο εισήγαγε διάφορα νέα στοιχεία στην αρχική πρόταση, όπως πιο ε, ε, φιλόδοξους στόχους, 20% για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων, την εισαγωγή του 7 της 7 πρόκλησης για θέματα κοινωνίας, για την ασφάλεια και επίσης προσπαθεί να διευρύνει τη συμμετοχή. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η συγγήτριά σας, Ρέαρα Μαντουρέλ, συμμερίζεται πολλές από τις ανησυχίες που εξέφρασε και το Συμβούλιο στην πρότασή του για τον κανονισμό πλαίσιο. Σημειώνουμε τη θετική προδιάθεση του Κοινοβουλίου για να αυξηθεί ο προπολογισμό Αναπόφευκτα το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τι συζητήσει για το πτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. σω το πιο σημαντικό νομοθετικό θέμα ενώπιον μα είναι οι κανόνε συμμετοχή και διάδοση του προγράμματο αυτού. Η Προεδρία μα θα επικεντρωθεί πολύ στου ε, δύο κανονισμού και κυρίω ε, στον κανονισμό για τη συμμετοχή. Και θέλουμε κυρίως να απλοποιήσουμε μέσω αυτού του κανονισμού. Αυτό το αίτημα προκύπτει εξελικτικά εδώ και μια σειρά ετών και χαίρομαι που οι διάφοροι εμπλεκόμενοι καλούν για αυτή την απλοποίηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως αναφέρεται στην έκθεση της κυρίας Καρβάλιου. Πρωταρχικός στόχος μιας τέτοιας απλοποίησης είναι πρώτον η μείωση του γραφειοκρατικού κόστους για τους συμμετέχοντες, η μείωση του χρόνου χορήγησης ε, επιδότησης και η μείωση του ενδεχομένου οικονομικών λαθών. Πρέπει βεβαίως να διατηρήσουμε την λεπτή ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνη και ελέγχου. Γι' αυτό η Επιτροπή προτείνει ένα σφαιρικό πρόγραμμα δέσμης απλοποίηση. Το συζητάμε και ω νομοθετική αρχή και με τους εμπλεκόμενου. Η συγκίτρια, ο εισηγητής ο κύριος Έκλερ, Πρόσφατα υπέβαλε το σχέδιο έκθεσης για τους κανόνες συμμετοχής. Οι συστάσεις του πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα. Πρέπει να συντονιστεί καλά η αντιμετώπιση του, λαμβάνοντας υπόψη τους στενούς δεσμούς μεταξύ των κανόνων συμμετοχής με τον ανθερμένο δυσμονικό κανονισμό και της κατεξουσιοδότησης πράξης. Η Προεδρία μας καταλαβαίνει τη σημασία απλοποιημένων και ευέλικτων κανόνων συμμετοχής για ένα επιτυχές πρόγραμμα ορίζον 2020 που θα διευκολύνει τη συμμετοχή των διαφόρων εμπλεκομένων και διασφαλίζοντας έτσι επαρκή επίπτωση του προγράμματος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Στόχος της Προεδρίας μας για το θέμα αυτό είναι να υπάρξουν έντονες συζητήσεις στο Συμβούλιο τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο με στόχο να καταλήξουμε σε γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια των ατύπων συναντήσεων, τη άτυπη συνάντηση των Υπουργών Έρευνα την επόμενη εβδομάδα στη Λευκοσία, θα κάνουμε ανταλλαγή απόψε για το θέμα αυτό και για τα πρότυπα χρηματοδότηση για την έρευνα για να διευκολύνουμε τη διαδικασία και ίσω να ανοίξουμε το δρόμο για τη συμφωνία στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι ένα τμήμα του, προγράμματος, του Γενικού Προγράμματος Πλαισίου για τις δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του ορίζοντα 2020 καθώς και τις συγκεκριμένες πλευρές εφαρμογής των διαφόρων δραστηριοτήτων. Εδώ με, με ενδιαφέρον παρατηρήσαμε τις διάφορες ε, προτάσεις της συγκήτρες κυρίας Καρβάλιου και προσβλέπουμε στην ε, γνωμοδότησή σας τον, ε, το φθινόπωρο. Θα είναι σημαντικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων Στόχος μας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι να επιτύχουμε μια μερική γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα το Δεκέμβριο. Και τέλος, έχουμε στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 ο κανονισμός πλαίσιο για το Ευρατόμ. Βεβαίως είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτό. Γιατί υπάρχουν ε, εκκλήσεις ε, επαναπροσανατολισμού για περισσότερη ασφάλεια και τον συνδυασμό με το πρόγραμμα ITER και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είμαστε ε, επιφυλακτικά αισιόδοξοι και θα επιδιώξουμε να υπάρξει μια μερική γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα το Δεκέμβριο. Ιδιαίτερα θα δώσουμε προσοχή στι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και προσβλέπουμε στη γνωμοδότηση τη Επιτροπή σα το φθινόπωρο. Δεύτερη προτεραιότητά μα είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία και Καινοτομία που προτάθηκε ως τμήμα του ορίζοντα 2020 για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Θεωρείται ότι θα συμβάλλει σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συνδυάζοντας και τις τρεις πλευρές του τριγώνου της γνώσης. Ιδιαίτερα ε, ασχολούμενο με την εκπαίδευση. Η πρώτη αξιολόγηση του Ινστιτούτου αυτού δείχνει σημαντική υποστήριξη στην ανάγκη ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, συνδυάζοντας την κορυφαία έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία σε, κοινότητε γνώση και καινοτομία, τα γνωστά KICS. Επίση, τα πορίσματα δείχνουν ότι υπάρχει ένα σαφέ δυναμικό και πολλέ ευκαιρίε για την μελλοντική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου. Όπω και ο δικό σου ηγετή, ο κ. Λάμπερτ και η κ. Τίερ και το Συμβούλιο, διαπίστωσε την ανάγκη για μια πιο ενδελεχή εξέταση των προτάσεων, όπως ε, το μοντέλο διακυβέρνησης, την επιλογή των νέων κοινοτήτων γνώση και καινοτομία και τι συνέργειε με τον ορίζοντα 2000. Επιπλέον, οι συζητήσει για τι νέε κοινότητε γνώση και καινοτομία συνδέεται άρρηκτα με τι συζητήσει για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Φυσικά θα λάβουμε υπόψη αυτή την αλληλεπίδραση και θα ε, πράξουμε τα δέοντα κατά την ε, συζήτηση της περαιτέρω από τον Κοινοτήτο Γνώση και καινοτομία. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μερική γενική προσέγγιση και για τα δύο θέματα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Θα ασχοληθούμε με τον κανονισμό του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Καινοτομίας τον Οκτώβριο και με το το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομία το Δεκέμβριο βάσει τη ε, διάσκεψη τη Κυπριακή Προεδρία που θα γίνει στην Κύπρο στι 8 και 9 Νοεμβρίου. Τρίτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι περίπου 95% τη έρευνα και τη καινοτομία και τη σχετική χρηματοδότηση γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών. Η αντιμετώπιση θεμάτων όπως ε, η διεύρυνση της ε, διασυνοριακής συνεργασίας και το άνοιγμα των αγορών εργασίας για τους ερευνητές, το θέμα της ισότητας φύλων σε ό,τι αφορά την ε, διακίνηση των ερευνητών θα συμβάλλουν αναμφίβολα στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα. Η Κυπριακή Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την μεγάλη επίβολη ιδέα ε, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα και προ τούτο θα συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα στην ε, ημερήσια διάταξη και των δύο Υπουργικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητα. Θεωρούμε ότι η διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε όχι μόνο ευκαιρίε, αλλά και προκλήσει και αυτό και η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα είναι μία από αυτέ. Ε, είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά και διαπιστώνω και τις σοβαρές ανησυχίες μερικών χωρών σε ό,τι αφορά τις γερικές ανισορροπίες και τη διείσδυση των διαφόρων προγραμμάτων. Η συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας θα ε, ε, προωθηθεί και από την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανανέεται την επόμενη εβδομάδα. προβλέπουμε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Οκτωβρίου όπου θα συζητήσουμε ταυτόχρονα και τα συμπεράσματα μιας συνδιάσκεψης του ΕΡΑ που θα γίνει στην Κύπρο στις 14 Νοεμβρίου. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα αυτό θα υιοθετηθούν στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τέταρτη και τελευταία μας προτεραιότητα είναι η πρόθεση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, έρευνα και καινοτομία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου. Είναι ευπρόσδεκτη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιλάβει την συνεργασία σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας με τις τρίτες χώρες προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του ορίζοντα 2020. Η Προεδρία μας πιστεύει ακράδαντα ότι το θέμα της διεθνούς συνεργασίας θα πρέπει να περιληφθεί οριζόντια σε όλα τα μέτρα για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και τους μηχανισμούς του ορίζοντα 2020. Και από αυτή την άποψη ε, περιμένουμε με αδημονία την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φθινοπόρου που θα συζητήσουμε το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο. Ένα άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Έρευνα στι 20 Ιουλίου θα εξετάσει τι διάφορε εναλλακτικέ λύσει και τι ευκαιρίε που προκύπτουν από την διεθνή συνεργασία με ιδιαίτερη έμφαση στην ε, ευρωμεσογειακή συνεργασία που μα είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Η έρευνα και η καινοτομία παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες ε, στις ε, μεσογειακές χώρες για να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους ε, αναπτύσσοντας τις οικονομίες τους. Και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μιας πολιτικής αστάθειας στην, περιοχή, στην ευρωμεσογειακή περιοχή, η πρόθεση πρωτοβουλειών για την έρευνα και την καινοτομία θα συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της κατάστασης στους ε, εταίρους μας της Μεσογείου και θα προλιάνουν το έδαφος προς μια οικονομική ανάπτυξη και μια πολιτική οριμότητα της περιοχής. Με βάση τη διακήρυξη και του Καΐρου το 2007 και αξιοποιώντας ε, τα πορίσματα της ε, Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης για την καινοτομία που έγινε στη Βαρκελόνη τον Απρίλιο θα συζητήσουμε και με τους υπουργούς ε, τέτοια είδους περιφερειακά προγράμματα καινοτομία που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων μας και ίσως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μία πρωτοβουλία στα πλαίσια του άρθρου 185. Θα το συζητήσουμε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα στι επόμενε εβδομάδε. Κυρία Πρόεδρε, εξότιμη Ευρωβουλευτέ, εν γνωρίζουμε ότι μία ομαλή μετάβαση από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στον ορίζοντα 2020 θα αποτελέσει ε, σημαντικό όφελος και για τους Ευρωπαίους ερευνητές και για την ευρωπαϊκή οικονομία και για να το καταφέρουμε θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Δυστυχώ ο χρόνο δεν είναι με το πλευρό μα. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρουν όσο το δυνατό πιο πολλά κοινά σημεία γίνονται του επόμενου μήνε προκειμένου να προλιάνουν το έδαφο και να διευκολύνουν την υλοποίηση συμφωνία φέτο. Είμαι πεπισμένο Πάντω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστερνίζεται αυτό το στόχο και προσβλέπω σε αγαστή και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ μα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μία επιφύλαξη. Οι προκλήσει ενώπιών μα δεν είναι μόνο να πείσουμε του ευρωπαίου πολίτε ότι εννοούμε αυτά που λέμε και ότι οι, πολιτικοί μας, οι πολιτικές μας όντως θα καταλήξουν στον στην πολυπόθετη οικονομική ανάπτυξη. Το βασικό δόγμα τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στηρίζεται στην ελληνική και στην άμυλα με την αξιοποίηση των καλύτερων πρακτικών. Οπότε να και στον καθένα από εμά να παραμείνει δεσμευμένος και προσιλωμένος στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και άσχετα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να συσπηρωθούμε να ε, τις υπερκεράσουμε έχοντας υπόψη αυτή την ε, βασική και πρωταρχική αρχή της αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την παρέμβασή σας. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ε, ντε καταρχήν. Έχετε το λόγο κύριε Κορέα Κάμπος. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μαλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την σαφέστατη εισήγησή σας και σας ευχαριστούμε γιατί παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας και δεσμευτήκατε για την ε, ταχεία έγκριση, που δεν θα είναι εύκολη, ε, έγκριση του ορίζοντα 2020. Αυτή είναι η άμεση προτεραιότητα της Επιτροπής μας επί του θέματος. Νομίζω ότι οι σχέσεις μας θα είναι πολύ καλές κατά το εξάμεινο της Κυπριακής Προεδρίας. Τρεις ερωτήσεις θα ήθελα να υποβάλω και είναι οι εξής. Εμείς έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Θεωρούμε ότι το EIT ίσως δεν περιλαμβάνει όλες τις ε, φιλόδοξες προβλέψεις του, αρχικές προβλέψεις τουλάχιστον και θεωρούσαμε ότι θα υπήρχαν υψηλές χρηματοδοτήσεις για το EIT Μας είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας είναι μία από τις προτεραιότητές σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο και εσείς έχετε αυτό το βασικό μέλημα και σας απασχολεί πραγματικά. Μας μιλήσατε για συγκεκριμένες υποδείξεις έτσι ώστε οι μικρομεσαίες χώρες να διαθέτουν περισσότερους πόρους στα πλαίσια της έρευνας, μέσα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Το θέμα αυτό δεν έχει επιληθεί δυστυχώς. Υπάρχει μεγάλος συγκεντρωτισμός πόρων μέχρι τούδε. Αυτό αφορά μία πολιτική η οποία δεν διέπεται πάντα από κίνητρα. Άρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ως προς την πολιτική συνοχής και την πιθανή χρήση των πόρων για να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και να μπορέσουμε να προωθήσουμε την επιστήμη και την καινοτομία. Τα προγράμματα αυτά είναι ευπρόσδεκτα για χώρες που δεν έχουν πρόβλημα υποδομών και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια για να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Έγινε λόγο στην Επιτροπή Περιφερειών και στο Κοινοβούλιο για το ότι ίσως ε, υπάρχει μία παρέκκληση ως προς τις περιφερειακές, ε, ε, την περιφερειακή προσέγγιση και την πολιτική χωρίς αποκλεισμούς. Πώς βλέπετε εσείς με τη συνεργασία, ε, πώς βλέπετε τη συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Θα ήθελα τη γνώμη σας και σε αυτό το σκέλος του ζητήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχω ερώτηση. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για πολύ απευθείας, ε, πάρα πολύ καλής ποιότητας και φιλόδοξη ομιλία μεταξύ όλων όσων έχω ακούσει. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να σε ευχηθώ ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και προσβλέπω πάρα πολύ στη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο Ρόντε. Ο κύριος Τζόνσον έχει το λόγο. Eh, Ο κύριος Γιώχανσον έχει το λόγο και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου ως προς τις ευχαριστίες ε, προς εσάς σε σχέση με τα σχέδια της Προεδρίας και τα σχόλιά σας προωθούμε και εμείς το πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων θα ήθελα και εγώ να ανταλλάξουμε απόψεις και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε θέματα επιστήμης πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Επίσης τι γίνεται με τη συνεργασία της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης. Εγώ ήμουνα επικεφαλής της ομάδας κατά την συνάντηση, τη διάσκεψη της Βαρκελόνης και θεωρούμε από πλευρά Σουηδίας ότι θα ήταν σκόπιμο να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία. Την είχαμε προωθήσει και στην περιοχή της Βαλτικής και μπορέσαμε να προχωρήσουμε αρκετά με χώρες που τώρα είναι κράτη-μέλη, αλλά δεν ήταν τότε. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τη συνεργασία με χώρες εκτός των συνόρων μας. Θα πρέπει να προωθήσουμε ανταλλαγές απόψεων και να μάθουμε πολλά, να αντιλήσουμε πολλά διδάγματα ημένα από τους δε. Είμαι υπέρ της συνεργασίας στην Μεσογειακή Λεκάνη. Ως προς τον ε, ορίζοντα 2020, εσείς ε, ε, μιλήσατε για τους συμμετοχικούς κανόνες. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που θα σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας υπέβαλα τροπολογίες. Είπα ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τους συμμετοχικούς κανόνες, υπάρχουν εισηγητές, υπάρχουν μέλη. Ας αρχίσουμε από αυτούς τους κανόνες συμμετοχής και ας δούμε και όλες τις ε, διακλαδώσεις που διαγράφονται πολλές φορές. Πρέπει να κινηθούμε στην πράξη και να απομακρύνουμε πρότυπα. Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας θα λάβουν το λόγο ακαδημαϊκοί και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε τους κανόνες συμμετοχής. Άρα προσβλέπω σε μια αγαστή συνεργασία μαζί σας και ελπίζω να ασχοληθούμε με τους συμμετοχικούς κανόνες. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε και με το δημοσιονομικό ζήτημα για τον ορίζοντα 2020. Μίλησατε για προκλήσεις και τις προκλήσεις που διαγράφονται ως προς την έρευνα, την βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός επί της δικής σας προεδρίας, αλλά θα πρέπει να τον προετοιμάσετε. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε σαφώς εγγεγραμμένες προτεραιότητες ποιες συζητήσεις θα προωθήσετε κατά την Προεδρία σας έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια πλειοψηφία στο Συμβούλιο και να προβούμε και σε επανακατανομή ε, δαπανών μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Ως προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ε, μιλάμε για αύξηση του προϋπολογισμού για το EIT. Εργάστηκα επί του θέματος και γνωρίζω ότι υπάρχει η υποστήριξη της βιομηχανίας, ε, τα ΚΙΚΣ, οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας μας υποστηρίζουν και ούτω καθεξής και ίσως οι έξι κοινότητες γνώσης θα πρέπει να τεθούν σε οριζόντιο επίπεδο, να υπάρχει μια οριζόντια προσέγγιση. Ποια είναι η άποψή σας για τα ΚΙΚΣ και την έξπος εποπτεία που προβλέπετε αυτών των μέσων. Ο κ. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ τον Κυπριών Υπουργών τον κύριο Σταύρο Μαλά στη συνεδρία μας. Να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ εμπεριστατωμένη και λεπτομερή παρουσίαση των θέσεων της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και να ευχηθώ στον ίδιο και στην Κυπριακή Προεδρία γενικότερα να αποδώσει τα μέγιστα έτσι ώστε στο τέλος αυτής της εξαμηνίας να φανεί ξεκάθαρα ότι η Κύπρος ε, δημιούργησε μια εικόνα πάρα πολύ θετική στον τομέα της ε, προεδρεύουσας χώρας. Έχω μια-δυο ε, ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ξεκινά με έναν προϋπολογισμό γύρω στα 80 δις. Αυτό όμως κατανέμεται μέσα σε μια περίοδο 6 χρόνων. Από αυτά τα 31,7 δις αναμένονται να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως αναγράφεται στην ίδια την πρόταση υγεία, ασφάλεια τροφίμων, αηφόρος γεωργία κλπ. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι μένουν περίπου 5,2 δις τον χρόνο για όλα τα κράτη, ποσό ελάχιστον μπροστά στον προϋπολογισμό βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι υπάρχουν τρόποι να αυξηθεί αυτό το ποσό και τι νομίζετε ότι μπορεί να επιτευχθεί από όσα α, ως πολύ ψηλούς στόχους έχετε θέσει εσείς μπορούν να υλοποιηθούν. Το δεύτερο ερώτημα, όταν πριν έξι μήνες επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Δανός Υπουργό Έρευνας και Κοινοτομίας, ο κύριος Σέστερ Γκάρτ, διαβεβαίωσε ότι η Δανέζικη Προεδρία θα δουλέψει για να διασφαλίσει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να επιτευχθεί μια γενική προσέγγιση στο Horizon 2020 μέχρι το Μάη του 2012 και να προχωρήσει η έναρξη του προγράμματος μέσα στο 2014. Αυτό έχει επιτευχθεί μερικώς. Ε, το ερώτημα είναι πώς σκοπεύει η Κυπριακή Προεδρία να προωθήσει το θέμα και προς ποια κατεύθυνση και θέλω να κλείσω με μια πιο γενική ερώτηση. Ε, κάθε ένας που αναλαμβάνει ένα μια υπεύθυνη αποστολή θέτει ασφαλώς συγκεκριμένους και ψηλούς στόχους. Το ερώτημα μου είναι με το τέλος αυτής της εξαμηνίας τι θα θέλατε εσείς οπωσδήποτε να μείνει ως έργο από όσα έχουν εξαγγελθεί. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι. Α, ο κύριος Μπουτικόφερ. Ευχα... Ευχαριστώ, ναι. Είχα ζητήσει το λόγο. Δύο ερωτήσεις. Είπατε ότι έχετε ελπίδες για να υπάρξει μία ομαλή μετάβαση από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 στον ορίζοντα 2020. Η ερώτηση μου είναι πώς θα γίνει αυτή η ομαλή μετάβαση στην πράξη πώς θα γίνει αυτή η ομαλή μετάγραφαση ούτως ώστε να είναι αποδοτική κιόλα, εάν το Συμβούλιο δεν δίνει τους αναγκαίους πόρους ούτε για να τηρήσουμε τις συμβατικές υποχρεώσει που έχουν συσσωρευτεί μέσα στο υπό το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μου πείτε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερη ερώτηση. Θα ήθελα την άποψή σας. για το πώς θα συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ορίζοντα 2020 και αυτό σχετίζεται και με τις παρατηρήσεις που έκανε ο Πορτογάλος συνάδελφος. Εδώ και πολύ καιρό συζητάμε για το ότι κάποιες ε, από τις χρηματοδοτήσεις μας, ένα ποσοστό πρέπει να πηγαίνουν αποκλειστικά στις μικρομεσαίες. Τι ποσοστό θέλετε εσείς, 0, 10, 20%. Στον ορίζοντα 20-20 τι ποσό πιστεύετε ότι πρέπει να πάει αποκλειστικά στις μικρομεσαίες και είστε διατεθειμένος να βοηθήσετε με ουσιαστική χρηματοδότηση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το εργαλείο για αυτές. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος δεν ζήτησε το λόγο, γι' αυτό δίνω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Ευχαριστώ για αυτό το ευρύ φάσμα ερωτήσεων και ιδιαίτερα φιλόδοξες ερωτήσεις, προκλητικές μάλλον. Ως προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και τις οικονομικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι επιστήμονες δεν τα έχουν καταφέρει τόσο καλά στην Ευρώπη, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολύπτυχη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του ακαδημαϊκού κόσμου της Ευρώπης είναι ότι δεν μπορεί να δελάσει, να προσελκύσει επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Οι ΥΠΑ τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα. Άρα το EIT ή οποιοδήποτε κοινό τεχνολογικό πρόγραμμα έρευνας θα πρέπει να προωθήσει αυτή την προσέγγιση, δηλαδή αυτή την πολιτισμική προσέγγιση προσέλκυσης επενδύσεων. Να υπάρχει μία επόαση δηλαδή αυτού του προγράμματος ε, συνέργειας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είχαμε τρεις ε, κοινότητες γνώσης, μιλούσαμε για 300 εκατομμύρια ευρώ αρχικά Και τώρα έχουμε ένα πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα. Θα δούμε κατά πόσο θα εξελιχθεί το πρόγραμμα για το EIT μέσα στα πλαίσια του πολιετούς προγράμματος. Θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Θα πρέπει να γίνει μία ενδιάμεση αναθεώρηση και να δούμε κατά πόσο η συμμετοχή της βιομηχανίας φτάνει σε ένα 75% όπως έχει προγραμματιστεί. Θα δούμε τι θα είναι, ποια θα είναι και τα πρώτα αποτελέσματα ως προς το σκέλος της εκπαίδευσης πρωταρχικά, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε καλύτερα ως προς την στρατηγική μας ατζέντα επενδύσεων ως προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, διότι θα λειτουργήσει συμπληρωματικά μέσα στα πλαίσια των καινοτομιών για τον ορίζοντα 2020. Άρα θα πρέπει να μιλήσουμε για συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, θα πρέπει να δούμε τις κοινέ τεχνολογίες και τον πυλώνα της εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια ενός συμπληρωματικού χαρακτήρα επενδύσεων ως προς τη βασική έρευνα. Και την κλίμακα θα την προσδιορίσουμε σε άμεση συνάρτηση με τον προϋπολογισμό. Ως προς την πρόσβαση, προσβασιμότητα, μιλούσατε για μικρομεσαίες χώρες, αν κατάλαβα καλά. Αυτό είναι ένα ουσιώδες ζήτημα και από εκεί και πέρα διακλαδίζεται η συζήτηση μέσα στα πλαίσια του προγράμματος έρευνας. Η Ευρώπη εμπλέκεται σε αυτή τη συζήτηση από το 2006. Έκτοτε γίνεται μία ολοένα και μεγαλύτερη συζήτηση κατά πόσο, για το κατά πόσο οι νέες χώρες στάθηκαν τόσο επιτυχής όσο είχαμε προβλέψει αρχικά. Ό,τι και να αποφασίσουμε θα βασιστούμε στην αριστεία και την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή με βάση την αριστεία. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και σημαίνει ότι θα πρέπει να προβούμε σε διαρθρωτικές αλλαγές για το πώς διενεργείται και προωθείται η έρευνα. Διατρέχουμε τον κίνδυνο μέσα στα πλαίσια της διευρυμένης ε, συμμετοχής να ολισθήσουμε από την αρχική συζήτηση και να φτάσουμε σε μια Ευρώπη δύο επιπέδων. Ως προς την πολιτική συνοχής, εδώ θα πρέπει να εμπλακούμε, διότι αυτό είναι το μέσο για τις μικρές και μεσαίες, μεσαίου μεγέθους χώρες, έτσι ώστε να προωθήσουν σχήματα αριστείας Δηλαδή τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορέσουν να συμμετάσχουν πιο εστιασμένα στις χώρες αυτές, μικρού και μεσαίου μεγέθους, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες τους, τα, σχήματα αριστείας για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα, προγράμματα έρευνας και ανταγωνισμού αρχικά αναφέρθηκα σε μία προειδοποίηση και η προειδοποίηση αφορούσε ακριβώς αυτό το σημείο. Ως προς τη συνεργασία με την Ανατολική Μεσόγειο, το θέμα αυτό έχει πολιτική πτυχή, μία πολιτική πτυχή, αλλά και μία οικονομική. Είμαστε γείτονες χώρες και εδώ διαγράφονται πολλές ευκαιρίες για οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Και εδώ μιλώ για εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Εδώ είχαμε μία επιτυχή διμερή συνεργασία με αυτές τις ε, χώρες της Βορείου Αφρικής Θέλουμε να επεκτείνουμε αυτό το σχήμα συνεργασίας. Μιλάμε για μια ουδέτερη πολιτική. Αυτό θα ακούσατε και στην αρχική μου δήλωση. Εδώ υπάρχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες μέσα στα πλαίσια των κλειδονισμών που γνωρίσαμε. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό, θα ήταν ένας παραγωγικός ε, παρεμβατισμός. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουτικόφερ για τα σχόλιά του. Κύριε Γιώχανσεν, νομίζω ότι ε, κάλυψα, σας κάλυψα με την απάντησή μου. Τώρα, οι συμμετοχικοί κανόνες, οι κανόνες συμμετοχής. Αυτό είναι το πιο, το, το πιο δυσχερές ζήτημα φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να λάβουμε στεναρές αποφάσεις. Στους κανόνες συμμετοχής υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά και τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε μιλήσει για πολλά σχήματα χρηματοδότησης των κανόνων συμμετοχής εσείς μιλήσατε για έναν εμπεριεκτικό κανόνα συμμετοχής που διέπει τα πάντα δηλαδή. Και θα πρέπει να το δούμε και από την οπτική γωνία των δικαιούχων. Εκεί ίσως πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις. Το είδαμε στο έκτο και το έβδομο πρόγραμμα ε, πλαίσιο. Εδώ έχουν οριστεί ε, διάφορα πρότυπα και μοντέλα. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν δούμε το πρόγραμμα υπαριθμών 5, το πλαίσιο ήταν πιο απλουστευμένο και η ζωή μας ευκολότερη. Γι' αυτό θα πρέπει να αντλήσουμε και ε, διδάγματα από το παρελθόν. Ως προς το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, δύο βουλευτές θίξατε αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω το συνολικό κόστος του ορίζοντα 2020, δεν εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιό μου. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο ζητά αύξηση του προϋπολογισμού αυτή η τάση διαγράφεται σε σχέση με το παρελθόν, όπου δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το συνολικό πακέτο και τι κονδύλια θα εμπεριέχει ο ορίζοντας 2020. Σας είπα ότι είναι φιλόδοξο το πρόγραμμά μας στην στρατηγική 2020 και επίσης σας είπα ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα περιεχόμενο σε αυτά που λέμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Μιλάμε λοιπόν για αυτό τον εμπεριεκτικό κανόνα και θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα φτάσουμε ως προς τον ορίζοντα 2020 και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό ε, Ινστιτούτο Τεχνολογίας και τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, τα ΚΙΚΣ νομίζω ότι σας κάλυψα. Ε, έχουμε να κάνουμε με τη μεγάλη εικόνα και τη μικρή εικόνα. Και εμβόλυμος μπαίνει φυσικά ο προϋπολογισμός. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μία μέση οδό που θα μας βρει όλους σύμφωνους. Κύριε Χατζηγεωργίου, ε, Νομίζω ότι σα σας κάλυψε όσον αφορά τον προπολογισμό στην απάντησή μου. Η Κυπριακή Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί να σφραγίσει όπως μας καλέσατε να σας πούμε πώς θα σφραγίσουμε τι σφραγίδα θα αφήσουμε θα προσπαθήσουμε να σε συμφωνία σε ένα-δύο θέματα σε αυτό το τομέα, γιατί ε, ο χρόνος μας λύγει. Πρέπει να ξεκινήσει το 2013 το πρόγραμμα αυτό. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να επιτύχουμε είναι κάτι συγκεκριμένο για τους κανόνες συμμετοχής. Είναι θέμα κλειδί. Πρέπει να είμαστε αρκετά πιο συμβιβαστικοί, να κατανοήσουμε τις θέσεις των άλλων διότι η συζήτηση ε, γίνεται όλο και πιο ταραχώδης. Να αποφύγουμε τον κίνδυνο να υπάρξει ένα σύστημα δύο επιπέδων, μια Ευρώπη δύο επιπέδων για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε λόγω της πολιτικής πίεσης, που αυξάνεται για το θέμα αυτό. Ο κύριος Μπιτικόφαρ ανέφερε κάτι πολύ σημαντικό πώς θα υπάρξει ομαλή μετάβαση από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 στον ορίζοντα 2020 εάν το Συμβούλιο σταματήσει, όπως έχει σταματήσει από ό,τι είπατε, αν κατάλαβα καλά, την χρηματοδότηση του τελευταί, της τελευταίας δέσμης προγραμμάτων. Όντως, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στη Δανία, εκφράστηκα πολύ κατηγορηματικά για το θέμα αυτό. Διότι στέλνουμε το πιο αρνητικό μήνυμα που θα μπορούσε κανείς να στείλει σε αυτή τη συγκυρία εάν δεν αποδεσμεύσουμε τις πληρωμές για τα προγράμματα αυτά. Και συμφωνώ μαζί σας ότι αν είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε, αν εννοούμε αυτά που λέμε, θα πρέπει οι πράξεις μας να είναι αντίστοιχες των λόγων μας. Καταλαβαίνω ότι κάποιες χώρες ε, αντιμετωπίζουν τις χέρειες. και ελπίζω να μην ε, θεωρούν ε, ότι η έρευνα δεν πρέπει πια να είναι προτεραιότητά τους, αλλά έχουν κάποιες χώρες δυσχέρειες που ίσως τις θέτει σε αυτή τη δυσχερή κατάσταση λοιπόν. Συμμετοχή των μικρομέσαιων επιχειρήσεων. Η ουσία είναι 20%. Αυτό θέλουμε εμείς αυτή τη στιγμή, το υποστηρίζουμε. Στο παρελθόν το επιτύχαμε, Κάναμε διάφορα πειράματα για τον τρόπο συμμετοχής των μικρομεσαίων στο παρελθόν. Κάναμε ταχυδεκτυλουργίες με τα νούμερα για να φτάσουν στο 15% που ήταν ο στόχος ε, του 7ου προγράμματος πλαισίου. Και τι εννοώ όταν μιλάω για ταχυδακτηλουργίες. Βεβαίως ε, ο βασικός μας στόχος ήταν 15% αλλά όταν περνάγαμε μετά στην εφαρμογή ε, προσπαθούσαμε να επιτύχουμε τα νούμερα και αν ε, δεν το επιτυχάναμε κάναμε κάποια υπολογιστικά κόλπα για να το επιτύχουμε στα χαρτιά. Έχουμε προγράμματα που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μικρομεσαίων για να φτάσουμε στο 20%. Και αυτό αυτή μας τώρα η προσέγγιση είναι από ε, ευθύ εξ αρχής πρέπει να επιδιώκουμε να φτάνουμε αυτό το 20% και όχι λογιστικά να το επιτυχάνουμε στο τέλος με κόλπα. Πάντα ήταν ατμομηχανή της ανάπτυξης μικρομεσαίες επιχείρησης στην Ευρώπη, πρέπει να τις υποστηρίξουμε όπως τις υποστηρίζαμε όπως τις υποστηρίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί μόνο οι μικρομεσαίες μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση. Είπα νωρίτερα για τις ε, κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, το EIT. Αυτή είναι η κόμβη όπου θα έπρεπε να προσπαθήσουν να κολλήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτοί είναι οι πυλώνες, αυτά είναι τα μέσα που, από όπου προκύπτει περισσότερη προστιθέμενη αξία η προστιθέμενη αξία ε, προκύπτει και επειδή συνεργάζονται με μεγάλες επιχειρήσεις και υπάρχουν έτσι διμερείς συνεργασίες, αλλά η έρευνα που κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο είναι πιο κοντά στις εφαρμογές, στην αγορά. Και αυτό χρειάζονται. θα ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην έρευνα και την αξιοποίηση της στην αγορά. Και για να γίνει αυτή η μετάβαση από το ένα στο άλλο πρέπει να υπάρξουν στρατηγικές πρωτοβουλίες και αυτές οι δημόσιες δυτικές πρωτοβουλίες είναι αυτές με τις οποίες θα μπορέσουμε να εμπλέξουμε περισσότερες μικρομεσαίες. Ευχαριστώ και να απάντησα σε όλα. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Διεξοδική ήταν η συζήτηση και άκρος ενδιαφέρουσα με την παρουσίασή σας και τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος της Επιτροπής και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι θα συνεδριάσουμε στις 3 το απόγευμα. Θα βρεθούμε εδώ εκείνη την ώρα στις 3 το απόγευμα. Γεια σας.